Good morning, ladies and gentlemen. Do you think we can begin our meeting for today? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω πως μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη σημερινή μας συνεδρίαση. Thank you. Thank you. Καλώς. Ε, ξεκινούμε λοιπόν με την ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, της 7ης Δεκεμβρίου του 2017. Ξεκινούμε λοιπόν με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν σχόλια σε σχέση με την ημερήσια διάταξη, προτάσεις, κύριε Βανίστελ Ρόι. Σας ευχαριστώ πολύ. Απλώς η Προεδρία δεν πρέπει να συνεχίζεται δύο φορέ. Ε, με την επερχόμενη Προεδρία δηλαδή. Ε, δεν έρχεται δηλαδή ο υπουργό εδώ στο πλαίσιο ακριβώ τη νέα ε, Προεδρία για να μα πει τι σκοπεύει να κάνει η νέα Προεδρία σε σχέση με την πολιτική συνοχή και επίση να μα ενημερώσει προηγούμενο προ τα αποτελέσματα. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο πλέον. Να λαμβάνουμε μια τέτοια ενημέρωση από τι Προεδρίε του Συμβουλίου. Δηλαδή κατά την έναρξη της θητείας τους και κατά το τέλος της θητείας τους έρχονται. Ε, δεν βλέπουμε όμως ε, στον νέο Υπουργό να παρευρίσκεται. Πρόεδρος, ε, ναι, δεν έχει προβλεφθεί συμμετοχή στη σημερινή συνεδρίαση. Ναι, θα γίνει μια συζήτηση τον Ιανουάριο με τη Νέα Προεδρία, αλλά αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ναι και πράγματι δεν έχουμε εδώ μαζί μας έναν στον Υπουργό. We, we had the meeting with him. Κατά την ε, διακοινοβουλευτική συνεδρίαση, δηλαδή με τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, κάναμε μια συζήτηση με τον Υπουργό. Παρευρέθηκε δηλαδή εκεί, στη συνεδρίαση της Επιτροπής ΡΕΓΚΙ, το Νοέμβριο με τα Εθνικά Κοινοβούλια και μας παρουσίασε τα επιτεύγματα της Εστονικής ε, Προεδρίας κάτι θητεία του. Οπότε παρευρέθηκε ναι στη συνεδρίασή μας. Υπάρχουν άλλα σχόλια σε σχέση με την ημερήσια διάταξη. Αν όχι, θεωρούμε πώ εγκρίνεται η μερίσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασης. Τώρα περνάμε στην έγκριση των ε, πρακτικών της συνεδρίασης της 13 η Νοεμβρίου. Ε, τα πρακτικά αυτά είναι διαθέσιμα online και ως συνήθως σας προτείνω πως εάν δεν υπάρχουν αστάσεις ε, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίας θα θεωρηθούν ως αγκεκριμένα ε, αυτά τα πρακτικά. Περνάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης της ανακοινώση της Προέδρου. Ε, έχω μία σειρά από ενημερωτικά σημεία από την πλευρά μου ε, για να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής. Καταρχήν, την, αυτήν τη Δευτέρα έγινε μία συνεδρίαση μεταξύ των τον Προέδρο των Επιτροπών και τον κύριο Σάντσεφ, ο οποίος είναι ο μόνιος αντιπρόσωπος ε, της Βουλγαρίας εδώ και, και είναι αρμόδιος για τα σχετικά ε, για τους σχετικούς νομοθετικούς εφακέλους και κατά συνέπεια θα χρειαστεί να συνεργαστούμε μαζί του κατά τους επόμενους ε, έξι μήνες και κυρίως στη συζήτησή μας εστιάσαμε στο πακέτο Omnibus το οποίο όμως ε, σκοπεύουμε να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τα τέλη του έτου, οπότε δεν νομίζω ότι θα εργαστούμε από αυτό με τη Βουλγαρική Προεδρία και μετά συζητήσαμε δύο ε, ακόμα φακέλους με τους οποίους, ε, επί των οποίων συμφωνήσαμε και έχουμε φτάσει σε μια προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο, αναμένοντας δηλαδή μια υπογραφή στο πλαίσιο της Ολομέλειας του Στρασβούργου και από εκεί και μετά αναφερθήκαμε Ε, στο γεγονός ότι στις 29 Μαΐου, τουλάχιστον αυτό μας είπε η Επιτροπή, θα υιοθετηθεί το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και από εκεί και μετά, πολύ σύντομα μετά από αυτό το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ενημερωθήκαμε ότι θα ακολουθήσουν νομοθετικές ε, προτάσεις. Δεν μας είπαν ακριβώς ε, πόσο γρήγορα, αλλά μας είπαν πολύ σύντομα μετά. Αυτό μας είπε η Επιτροπή και το Συμβούλιο. Επίσης, κάτι ακόμα για το οποίο μας ενημέρωσε η επερχόμενη Προεδρία είναι ότι θα διοργανώσει μια εμ, διάσκεψη κορυφής ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Πολιτική ε, Συνοχής και την τις προοπτικές μετά το 2020. Στη Σόφια λοιπόν θα λάβει χώρα τον Ιούνιο του 2018 και άτυπος, χωρίς δηλαδή να αποστείλω επίσημη επιστολή, ε, ζήτησα εκεί να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής μιας αντιπροσωπείας από την πλευρά της Επιτροπής Τώρα, στις 15 Νοεμβρίου, παρευρέθηκα σε μια διάσκεψη στο Στρασβούργο που διοργανώθηκε από τον Επιτρόπο σε ό,τι αφορά την επένδυση στη διασύνδεση της Ευρώπης και Ανάμεσα στα κυριότερα ζητήματα ε, που συζητήθηκαν ήταν το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, και ε, τα αποτελέσματα του, του προγράμματος διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, το Connected Europe Facility, το οποίο έχει πλήρως πλέον εκταμεθεί, δηλαδή στο 93% και το επίπεδο των, της φιλοδοξία μας σε σχέση με τις μελλοντικές επενδύσεις, τα μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα στις μεταφορές και υπήρξε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα ότι είναι απολύτω απαραίτητε οι επενδύσει στον τομέα των μεταφορών και κανεί δεν έχει αντίρρηση απέναντι σε αυτό. Αλλά το όραμα του Επιτρόπου είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη, αλλά όχι ε, χρηματοδότηση μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Και αυτό γιατί η εν λόγω διευκόλυνση τη χάνει καλύτερη διαχείριση, είναι πιο συγκεντρωμένη, πιο κεντρική και επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό ήταν δηλαδή το κύριο ε, μήνυμα που προέκυψε από αυτές τις συζητήσεις. Σε ό,τι αφορά το μελλοντικό MFF, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, από αυτή την πλευρά, από, αυτόν, από αυτούς δηλαδή που ενδιαφερόμαστε για τις μεταφορές, ήταν ότι ε, θα είναι η συνολική επένδυση μέσα σε αυτό το πλαίσιο 700 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, επόμενη ανακοίνωση που θα ήθελα να κάνω η, τελευταία πρωτοβουλία από την πλευρά της Επιτροπής. Ίσως τα ακούσατε δηλαδή ότι χθε το πρωί η Επιτροπή συζήτησε ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει και νομοθετικές προτάσεις αλλά και έγγραφα θέσεις, position papers για την επανεκκίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την οικονομική κρίση και σε συνέχεια της απόφασης ε, του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην επόμενη διάσκεψη κορυφή του Συμβουλίου, 14 και 15 ε, Δεκεμβρίου, θα γίνει σχετική συζήτηση. Δύο από αυτά τα ζητήματα αφορούσαν τη δική μας Επιτροπή και είχαν να κάνουν και τα δύο με τις διατροφικές μεταρρυθμίσεις. Το πρώτο από αυτά αφορά την αναθεώρηση ε, του κανονισμού σε ό,τι αφορά το Ταμείο για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων και οι προτάσει που έχουν γίνει εδώ περιλαμβάνουν ε, την αύξηση του σχετικού προπολογισμού από 143 εκατομμύρια ευρώ σε 300 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο από το 2017 στο 2020. Και επίσης ε, προτάθηκε ο στόχος του προγράμματος να στοχεύει περισσότερο στα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία προετοιμάζονται για προσχώρηση στην Ευρωζώνη. Ε, η δεύτερη από τις προτάσεις που μας αφορά είναι η τροποποίηση του ε, κανονισμού για τις κοινέ διατάξεις έτσι ώστε να επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αξιοποιούν το performance reserve όπως λέγεται στα υπάρχοντα ε, διαρθρωτικά ταμεία προκειμένου να υποστηρίζουν διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει αντί να ε, ε, στηρίζουν πολύ συγκεκριμένα project. Καθώ τα σχετικά αποθεματικά αντιστοιχούν στο 6% των σχετικών επιστώσεων στο πλαίσιο του ΕΦΣΥ, κάποια από αυτά τα κονδύλια είναι πολύ ψηλά, ως, δηλαδή σύνολο για κάθε κράτο μέλο. ανά κράτο μέλο, βέβαια αυτό. Διαφοροποιείται αυτό το ποσό. και αναμένω πως οι, οι εν λόγω προτάσεις θα ανακοινωθούν στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα. Και αναμένουμε πως βέβαια θα αναφερθεί η ΡΕΓΙ ως η αρμόδια επιτροπή για αυτούς τους φακέλους. Βέβαια το τι ακριβώς θα συζητηθεί εκεί θα τα ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα. Οπότε αναμένω εδώ και κάποια διαμάχια ανάμεσα στη δική μας επιτροπή και τις υπόλοιπες επιτροπές όπως είχε γίνει και ευθύ εξ αρχής ε, όταν άρχισε να συζητείται δηλαδή το πρόγραμμα για, τις, ε, για την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Ο κ. Βανίλιστερο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πληροφόρηση αυτή, για τις εργασίες το επόμενο εξάμεινο και τις επιπτώσεις στο MFF. Σε σχέση με το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη, το ΣΕΦ, καθίσταται σαφές ότι όταν μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Σύνοχης και τη συνεισφορά στο ΣΕΦ, καθίσταται σαφές ότι μιλάμε για στόχους συνοχής, για χρήματα συνοχής και καλύτερο μέσο δαπάνης. Έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη απόδοση. Ε, δεν ε, θέλω να φτάσω σε γρήγορα συμπεράσματα. Φυσικά τα χρήματα θα βρίσκονται στο ΣΕΦ. Και αυτό δεν αφορά ούτε τις αποφάσεις της Επιτροπής Μεταφορών, ούτε τις δικές μας. Γιατί φυσικά θέλουμε να έχουμε καλύτερες ε, διασυνοριακές λύσεις και αποδόσεις, αλλά θα πρέπει να εργαστούμε ε, επ' αυτού. Υπάρχει ε, μία έκθεση του κυρίου Νοβακόφ για την εφαρμογή του πλαισίου και θα πρέπει να συνδέσουμε τα δύο γιατί έχει μεγάλη σημασία να δούμε ποιες είναι οι απόψεις ως προς αυτή τη ε, ε, διασύνδεση σε σχέση με την χτεσινή πρόταση είναι ακριβώς αυτό που είχατε πει. Δηλαδή, αυτή η αλλαγή του κανονισμού που θα φτάσει στην Ολομέλεια, όπου έχουμε πολύ καλό έρισμα για τις περιφέρειες και τις πόλεις σε αυτό το πρόγραμμα στήριξης το οποίο λειτουργεί καλά σε σχέση με τις χώρες που το ζήτησαν. Το, ε, η πρώτη δόση του 2017 ήταν πολύ μεγάλη και τώρα βρέθηκαν επιπλέον χρήματα κάπου στο περιθώριο για την επέκταση αυτού του προγράμματος. Ο κανονισμός είναι δικός μας και αν αλλάξει ο κανονισμός η ΕΚΟΝ μπορεί να γνωμοδοτήσει, αλλά ο κανονισμός είναι δικός μας. Θα πρέπει να δώσουμε μάχη για να παραμείνει εδώ. Θα πρέπει να δούμε το MFF σε πρώτη φάση, γιατί δεν θα πρέπει να περάσει αυτή η αρμοδιότητα στην ΕΚΟΝ στη συνέχεια. Είναι μια κρίσιμη στιγμή, βρισκόμαστε σε μια καμπή και το ταχύτερο δυνατόν. Βασίζομαι σε εσά και στη γραμματεία. Μετά από τις πληροφορίες που θα λάβουμε την επόμενη εβδομάδα. Ίσως θα το συζητήσουμε αργότερα στους συντονιστές. Σας ευχαριστώ. Βεβαίως θα το δούμε με τους συντονιστές. Αλλά θα πρέπει να πω ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια, όπως και στην προηγούμενη περίσταση δεν ήταν καθόλου εύκολο και το ξέρετε αυτό, αλλά ε, μετά από την υποστήριξη των πολιτικών ομάδων καταφέραμε εμείς να είμαστε η υπεύθυνη, η αρμόδια καθήλυν επιτροπή, διότι κινηθήκαμε από κοινού. Ο κύριος ε, Ζέλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ε, κάποια, κάποια τμήματα της Επιτροπής τα οποία προσπαθήσουν να προωθήσουν τους δικούς τους ε, φακέλους, πράγμα το οποίο όμως αποβαίνει, αποβαίνει βάρος της περιφερειακής πολιτικής. Για παράδειγμα, στον τομέα της απασχόλησης θέλουν να ξεχωρίσουν, να, να, να διαχωριστεί το, υφιστάμενο ε, ταμείο και να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό ταμείο για την ε, ε, καταπολέμηση της απασχόλησης. Έτσι δηλαδή θα υπάρχει κάτι παράλληλο, μια παράλληλη προσπάθεια, ένα παράλληλο ταμείο προς την πολιτική συνοχή. Και από την πλευρά της, ε, των μεταφορών βλέπουμε κάτι αντίστοιχο στο πλαίσιο δηλαδή της ε, διευκόλυνσης συνδέοντα στην Ευρώπη. Οπότε νομίζω πως θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε το επόμενο διάστημα έτσι ώστε να συνεδριάσουμε από κοινό επιτροπές και να δούμε κατά πόσο επιθυμούμε ένα τέτοιο κατακαιρματισμό αν θέλετε της πολιτικής συνοχής. Ε, ειδικότερα ο τομέας των μεταφορών μου φαίνεται πως είναι πολύ σημαντικός γιατί το, το πρόγραμμα συνδέοντα στην Ευρώπη είναι τελείω διαφορετικό προ τη στοχοθεσία του. Δηλαδή, στοχεύει στο, ότι όταν στο διασυνοριακό, στη διασυνοριακή κυκλοφορία υπάρχουν προβλήματα, ε, υπάρχουν δηλαδή bottlenecks όπως λέγονται, σημεία συμφόρησης, ε, έχει στόχο στο να ε, επιλύονται αυτές οι συμφορήσεις. Αλλά εάν δούμε για παράδειγμα ποια είναι η κατάσταση των σιδηροδρόμων σήμερα στην Ευρώπη, δεν έχει επιτύχει τους στόχους του αυτό, το, αυτή η διευκόλυνση. Και τώρα ε, θέλουμε άλλα, άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, μη βλέπουμε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ε, η Κίνα, να ανοίξουν έτσι προγράμματα και οδούς μεταφορών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση Ε, και τέτοιου είδους βέβαια προσπάθειες που γίνονται από αυτές τις χώρες έρχονται σε αντίθεση ε, με όλες τις προσπάθειες δεκαετιών που έχουμε κάνει μέσω των ευρωπαϊκών ε, δικτύων μεταφορών. Θα πρέπει λοιπόν να επιτύχουμε εκείνα που πρέπει να επιτύχουμε, δηλαδή ε, βελτιώσει ειδικότερα στους σιδηροδρόμους, γιατί οι σιδηροδρόμοι παραμένουν τελικά σε μια κατάσταση όπου δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς. Ε, αντιθέτως έχουν υποκατασταθεί από το δικό δίκτυο. Ε, και ε, εδώ έχουν γίνει ε, πολλά από τα προβλήματα οφείλονται στα κράτη-μέλη τα οποία δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν μεταξύ τους ως προς το ποια λύση θα έπρεπε να βρεθεί. Ε, για παράδειγμα, δεν υπάρχει συνδρομική τη σήμερα ημέρα σύνδεση μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνία, γιατί το δίκτυο είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση που ούτε με 30 χιλιόμετρα ανά ώρα δεν μπορούν να κινούνται τα τρένα. Αυτό για μένα είναι σκανδαλώδε. Ε, άρα λοιπόν στο πλαίσιο ε, της τρέχουσας ε, προγραμματικής περίοδου βλέπετε κάτι τέτοιο, αλλά η κινητικότητα και τα μέσα μεταφοράς εντός των πόλεων θα έπρεπε να αποτελέσουν και αυτά προτεραιότητες. Οπότε όταν μας λένε τώρα ότι είναι ευκολότερο στη διαχείριση το πρόγραμμα διευκολύνσης της Ευρώπης, εντάξει δεν είμαι σίγουρος, θα πρέπει να το ελέγξουμε. Νομίζω δηλαδή πως ένα τμήμα των σχετικών κονδυλίων τελικά ε, βγήκε από τη διευκόλυνση της Ευρώπης για να χρηματοδοτηθεί το ΕΦΣΙ και τώρα ε, προσπαθούν ουσιαστικά να ε, και πάλι να συμπληρώσουν τα κονδύλια που χρειάζονται για άλλε προτεραιότητε από την πολιτική συνοχή, βγάζοντας τα από την πολιτική συνοχή. Και νομίζω πως θα πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα στιγμή με τους συναδέλφου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Κέλ. Έχει το λόγο. Ναι. Ε, θα υποστηρίξω ε, πλήρως τα όσα είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Δηλαδή, πρόκειται για μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά θέλει να μας δώσει ένα μήνυμα ότι θα πρέπει να βγουν χρήματα, να βγουν κοντήλια από την πολιτική συνοχή προτού εγκρίνουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, γιατί τελικά δεν θα φτάσουμε εκεί που χρειαζόμαστε σε ό,τι αφορά τα ε, κονδύλια. Και αυτό το αποθεματικό απόδοση, αυτό το performance reserve, είχαμε πει ότι δεν θέλουμε να αξιοποιηθεί και ε, είχαμε ε, πράγματι δίκιο. Όταν δηλαδή μας λέει η Επιτροπή ότι θέλει να το αξιοποιήσει με διαφορετικό τρόπο, δεν μπορούμε να το δεχτούμε όταν δηλαδή θα κατευθυνθεί προς ένα εργαλείο το οποίο δεν εμπίπτει στο δικό μας τομέα αρμοδιότητας. Και επίσης ε, ε δεν αντιλαμβάνομαι ε, εάν έχει ληφθεί μια απόφαση πέρα της παράτασης της ύπαρξης του SSP έως το 2020. Δηλαδή είχαμε πει ότι μέχρι τότε θα προβλέπεται μια υποστήριξη ως τεχνική υποστήριξη, αλλά από εκεί και μετά δεν ξέρω γιατί λέμε εκ των προτέρων ότι θέλουμε να περιληφθεί και στο επόμενο πολιτικό σε δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Ουσιαστικά δηλαδή αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις ε, για ένα τέτοιο πρόγραμμα πέραν του τρέχοντος ε, δημοσιονομικού πλαισίου δεν είναι κάτι τέτοιο ρηψοκίνδυνο. Θα πρέπει λοιπόν να περάσουμε ευθύτερα το μήνυμα ότι εμείς είμαστε αρμόδια επιτροπή και θα μείνουμε αρμόδια επιτροπή και ε, η επιτροπή θα πρέπει να μας δέσει πολύ ξεκάθαρες εξηγήσεις ως προς το γιατί πρέπει να υποστηρίξουμε αυτές τις προτάσεις που έχει κάνει. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λάβει απαραίτητες εξηγήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τις εξηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη ανέφερα και δύο φορές ότι καλέσαμε τον Επίτροπο Ντομπρόφσκης λόγω του τέλους της πρώτης φάσης του προγράμματος. Οπότε τον περιμένουμε τον Φεβρουάριο. Θα έρθει στην Επιτροπή μας. Βασικά θέλουμε να σχεδιάσουμε τα αποτελέσματα του προγράμματος. Αυτό θέλαμε. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε τα αποτελέσματα του προγράμματος και προτάσεις για παράταση του προγράμματος. Τελευταίος ομιλητής, διότι είμαστε ακόμα στις ανακοινώσεις του κ. Μποστινάρου. Ευχαριστώ. Δεν θα μακρηγορήσω. Σαν πρώην εισηγητής για το Ταμείο Συνοχής, θυμόμαστε όλοι ότι πιθανότατα ήταν η σημαντικότατη μάχη που δώσαμε την προηγούμενη φορά. Να πείσουμε ότι το μέσο για τη σύνδεση της Ευρώπης, το ΣΕΦ, δεν θα έπρεπε να είναι ένας τρόπος για να βγάλουμε χρήματα από τη συνοχή. Τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. χωρίς να δούμε μια αξιολόγηση πώς δαπανήθηκαν τα χρήματα. Γι' αυτό και εγώ υποστηρίζω την πρόταση Λάμπερτ. Πρέπει να ζητήσουμε μια αξιολόγηση. Πώς δαπανήθηκαν τα χρήματα. Επίσης, θα ήθελα λεπτομερέστατα αποτελέσματα περί γεωγραφικής κατανομής της χρήσης του ΣΕΦ κάθε κράτος μέλος πώς έχει πρόσβαση στα χρήματα του ΣΕΦ πόσα χρήματα μεταφέρθηκαν από πρώτη θα μεταφέρονται πρώτη πρώτου 2018 στις Βρυξέλλες και ποια είναι τα αποτελέσματα. Πού κάνει τη διαφορά το μέσο και τη διασύνδεση της Ευρώπης εν συγκρίση με, την, ε, το Ταμείο Συνοχής και πώς βελτιώνουμε δυσυνοριακά την διασυνδεσιμότητα. Πόσο βελτιώθηκε η κατάσταση, η ενέργεια, το φυσικό αέριο, οι βριζονικές υπηρεσίες, οι σιδεδρομικές ε, μεταφορές. Όχι ε, μόνο οι αυτοκινητόδρομοι. Χωρίς αξιολόγηση συνεπιών, εμείς πρέπει να είμαστε αντίθετοι όσον αφορά τη μεταφορά πόρων. Διότι, όπω είπε η Κωνσταντσέ, πρέπει να προσθέσουμε και άμυνα και μετανάστευση και ασφάλεια. Και μειώνεται το ποσό που έχουμε στην τσέπη μας με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου. Ολοκληρώνεται αυτή η μικρή συζήτηση που έλαβε χώρα στις ανακοινώσεις της Προέδρου και έχω να πω ότι θα συναντήσουμε την Επίτροπο Κρέτσο και νομίζω ότι θα πρέπει να στρέσουμε ένα σοβαρό θέμα και να υποβάλουμε σχετικό αίτημα. Όταν βλέπουμε τέτοιες επιθυμίες που εκφράζονται από διάφορες πολιτικές, κοινωνικές πολιτικές, μεταφορές, επιθυμίες περικοπών να αποσπαστούν χρήματα από την πολιτική συνοχής και να δημιουργούνται νέες προσεγγίσεις και πακέτα μέτρων, Πρέπει να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι η άποψη της Επιτροπής, του Αρμόδιου Επιτρόπου για την Περιφερειακή Πολιτική. Ποια είναι τα σχέδια του Επιτρόπου για Περιφερειακή Πολιτική πριν προταθεί το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Διότι εδώ προσπαθούμε στο Κοινοβούλιο προσπαθούμε να κινηθούμε μεταξύ δύο πραγμάτων. Θέλουμε καταρχάς να δούμε σημαντικά Θέλουμε μάλλον να δούμε μηνύματα ξεκάθαρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα κινηθεί. Ολοκληρώνουμε αυτό. Τελευταία ανακοίνωση. Άλλη κατεύθυνση ακολουθεί αυτή. Φέτος δεν θα έχουμε πάρτι για τα Χριστούγεννα. Έχουμε τόσες γιορτές για τα Χριστούγεννα. Τόσες πολλές εκδηλώσεις που δεν μπορούσαμε να βρούμε χώρο και χρόνο για το δικό μας πάρτι. Και εκείνοι που έχουν, ξέρουμε ότι δεν πηγαίνουν πολύ σε αυτά τα χριστουγεννιάτικα πάρτι στο Στρασβούργο. Έχουμε κακή εμπειρία. Γι' αυτό θα έχουμε ένα πάρτι για τον νέο χρόνο αμέσως μετά την πρώτη μας συνεδρίαση εδώ τον Ιανουάριο. Και ελπίζουμε να είναι μια καλή εκδήλωση, καλή ευκαιρία να ευχηθούμε ημέν τους δε, καλή επιτυχία και καλή διάθεση κλπ. Αυτή είναι η τελευταία μου ανακοίνωση και μπορούμε να συνεχίσουμε την ημερήσια διάταξη και πάμε στις ψηφοφορίες. Ψηφίζουμε τώρα λοιπόν τη γνωμοδότηση που ετοίμασε η κυρία Μόνικα Σμόλκοβα. Αφορά την ε, επιτροπή που φορά την επιτροπή πρόσβα, επιτάχυνση ε, της καινοτομία για καθαρότερη ενέργεια. Συνέταξε την γνωμοδότησή τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, 16 Οκτωβρίου ήταν η ημερομηνία τη τροπολογία, 63 τροπολογίες υπευλήθησαν. Και ε, η συγγήτρια προτείνει 12 συμβιβαστικές. Θα εγκριθεί η έκθεση τον ε, Ιανουάριο από την ε, αρμόδια επιτροπή. Η κυρία Σμόλκοβα θέλει να πει ορισμένα λόγια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την εργασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία και τους Σκιώδες και νομίζω θα έχουμε μια πολύ καλή έκθεση προς την ε, Ήτρε που θα δώσουμε στην Ήτρε. Αρχίζουμε με την ψηφοφορία. Τροπολογία 1 με συγχωρείτε, συμβιβαστική 1. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, λέει η Πρόεδρος, συμβαστική 2. Θα προσπαθήσω να συγκεντρωθώ. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε? Όχι. Δεν είμαστε στην Ολομέλεια. Ωραία, σας ευχαριστώ. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία η 18 καταπίπτει. Τροπολογία 22 καταπίπτει. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 56. Ψηφίζουμε την 56 υπέρ, κατά, αποχές, ας ελέγξουμε. Τροπολογία 56. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. And it is... εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 60. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Και τώρα, συμβιβαστική 12. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote Πέρας. Και εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Συγχαρητήρια κυρία Σμόλκοβα. Τώρα συνεχίζουμε. με την, ε, το προσχέδιο έκθεσης για τις περιφέρειες που έχουν μείνει πίσω. Είναι η ίδια πρωτοβουλία για τις περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Τζουφρίντα είναι η εισηγήτρη. Α, με συγχωρείτε. Σήμερα δεν είμαι και στα πολύ καλά μου. Δικό μου λάθος, πριν από το θέμα αυτό, για τις περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση έχουμε την ανταλλαγή απόψεων επί της έκθεσης Βαλίνα «Ο ρόλος των περιφερειών και πόλεων στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων, COP21». Η Ρέτζη έχει συντάξει η ίδια έκθεση και γνωμοδοτήσαμε στις 24 θα γνωμοδοτήσουμε στις 24 Δεκεμβρίου. Παρακαλώ να είσαστε λίγο πιο ήσυχοι. Εννοούσε 24 Νοεμβρίου η Πρόεδρος. Τώρα θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Κύριε Νοβακόφ, κύριε Μποστινάρο, να σας επαναφέρω στην τάξη. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια και θα ήθελα την προσοχή του κοινού. Κυρία Μολίνα, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ πολύ γιατί έχετε την έκθεση στη, στον ιστότοπό μας και νομίζω ότι την παρακολουθήσατε. Επίσης θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας απόψεις και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο δεν τα πηγαίνουμε και πολύ καλά. Έχουμε καθυστερήσει ιδιαίτερα σε σχέση με την εφαρμογή ε, διορθωτικών λύσεων, όπως συζητήσαμε και στο θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσπαθούμε να συλλέξουμε μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν σε επίπεδο πολιτικής συνοχής καθώς και περιφερειών. Οι κλιματικές αλλαγές καταδεικνύουν τις κοινωνικές διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε πιο ευαίσθητη θέση, διαφορά φύλου, χαμηλά εισοδήματα και ισότητες μεταξύ ανδρών και ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Ευρώπη φέρει μεγάλη ευθύνη για να απαλύνει τις ανθρωπιστικές συνέπειες που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Μιλάμε για ε, για ξηρασία και φυσικά και ένα μεγάλο κύμα προσφύγων που καταφεύγουν στην Ευρώπη εξαιτία των κλιματικών αλλαγών στις περιοχές τους. Ακριβώς γι' αυτό μιλήσαμε για την ανάγκη υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια δημιουργίας ε, πηγών πληροφόρησης καθώς και τεχνογνωσίας, χρηματοδότησης και επιστημονικών γνώσεων θα θέλαμε να επιμείνουμε για μια μεγαλύτερη αυτονόμηση των περιφερειών και των τοπικών φορέων. Γι' αυτό χρειάζονται μέτρα τα οποία δεν θα πρέπει να είναι πάντα υπερεθνικά. Μιλάμε για τις πόλεις και τις περιφέρειες. Αυτές είναι οι λέξεις ε, κλειδί οι τοπικές αρχές είναι αυτές που έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να απαντήσουν επαρκώς και έτσι ώστε οι πόλεις να καταπολεμήσουν τις κλιματικές αλλαγές. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουν πολιτική και οικονομική αυτονομία. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μέτρα αντιμετώπισης και εξομάλυνσης θα πρέπει επίσης να καταδικάσουμε την απόσυρση των ήπα από το σύμφωνο που αφορά την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών από την COP 21, 22, 23. Η απανθρακοποίηση επίσης θα πρέπει να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας έτσι ώστε να ενδυναμωθεί ο κοινωνικός ιστός. Έτσι θα χρησιμοποιήσουμε ανανεώσιμες περισσότερο, αλλά θα πρέπει επίσης να έχουμε και επενδυτικά σχέδια, καθώς και σχέδια αλλαγής δραστηριότητας μακροοικονομικά. Και επίσης αυτή η υποστήριξη θα πρέπει να φτάσει απευθείας στα νοικοκυριά που πλήττονται και όχι στις πολυεθνικές του τομέα της ενέργειας όπως συμβαίνει στη χώρα μου. Επίσης θα πρέπει να υπενθυμίσουμε τη γενεά των ανθρώπων που μετατρέπονται σε πρόσφυγες για λόγους κλιματικών αλλαγών και τις ε, που οδηγούν σε αυτό το μεγάλο προσφυγικό κύμα αυτό το θέμα φυσικά σχετίζεται και με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες που ε, καταφεύγουν στην Ευρώπη από τις ε, χώρες τους για λόγους κλιματικών αλλαγών αλλά και εμπόλεμων σειράξεων. Γι' αυτό θα πρέπει να εφαρμόσουμε και την πολιτική ισότητας μεταξύ των δύο φύλων κατά την εφαρμογή και αξιολόγηση των μέτρων καθώς και μία ενδελεχή ανάλυση όλων των τομέων που, και μέτρων που προτείνουμε. Τέλος, θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα κακού μάλλον προγραμματισμού και έλλειψη συντονισμού. Είναι ένα παράδειγμα, ένα απτό παράδειγμα το οποίο ζούμε. Θα έχετε λάβει μία ανακοίνωση για την επόμενο σύνοδο όσοι θα μεταβείτε οδικός και γνωρίζετε ότι θα πρέπει να ε, βάλετε μία ε, βινιέτα στο παρμπρίς για τις εκπομπές ε, καυσαερίων. Αυτό ισχύει στη Γερμανία εδώ και χρόνια και στη ε, είναι η Ισπανία σε ορισμένες πόλεις. Επίσης στην Αυστρία, Δανία και Τσεχική Δημοκρατία είναι υποχρεωτικό για μια σειρά οχημάτων. Εάν λοιπόν ε, υπάρχει η βινιέτα για τα τέλη κυκλοφορίας και για τον τεχνικό έλεγχο θα, ή ας πούμε για ε, να μπορέσουν να παρκάρουν εκεί που εργάζονται. Θα πρέπει επίσης ε, να λάβουμε υπόψη ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει και ειδική βινιέτα για τις εκπομπές καυσαερίων. Δηλαδή είναι πολύ καλές οι προθέσεις καταρχήν, αλλά δυστυχώς υπάρχει κάκιστος ε, προγραμματισμός και αποσυντονισμός. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε αυτό το πλαίσιο και είναι φυσικά ευπρόσδεκτες όλες οι υποδείξεις σας για τη βελτίωση αυτής της έκθεσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω στα μέλη το λόγο. Η πρώτα. Η κυρία Σπυράκη. Κάποια κάποιος μιλήσει εκ μέρους της κυρίας Σπυράκη. Ο κ. Βανίστερ Ρόι. Δεν ήρθα ακόμα. Άκουσα προσεκτικά και κατανοώ κάποια ισπανικά ακόμα. Σας παρακολουθώ στα ισπανικά. Αληθεύει ότι ο ρόλος των περιφερειών και των πόλεων ε, ε, βαίνει αυξανόμενος. Και κυρίως σε αυτό το τομέα του κλίματος και της ενέργειας και τους στόχους που έχουμε θέσει. Γι' αυτό δεν μιλάμε για νέους στόχους. Είναι αποδεκτή. Στο Παρίσι. Περισσότερο για επιδόσεις νοιαζόμαστε. Και όπως είπαμε και πριν από λίγα λεπτά, υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες στον τομέα μας. Έχουμε επιδόσεις που ε, και πολλά διαθέσιμα χρήματα. Ας είμαστε δημιουργικοί. Μέσω της εκθέσεως μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε, να βελτιώσουμε τις επιδόσεις με δημιουργικό τρόπο. Είπατε ότι έχουμε πολλά νέα μέσα για την ενεργειακή μετάβαση που αποδίδει η επένδυση και σε, μετά από 10 χρόνια. Μέσω εξοικονόμησης ενεργείας, αποδόσεως της ενέργειας, βιώσιμης ενέργειας επιστρέφουν τα χρήματα. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και διάφορα άλλα προγράμματα. που μπορούν να βοηθήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση, να επενδύσουν μαζί με τους εταίρους τους, να κάνουν τις επενδύσεις που θα αποσβεστούν αργότερα και θα αποδώσουν κέρδη. Και μπορούμε να επηρεάσουμε τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι πόλεις. Δεν είναι εδώ κυρία Σπυράκη. Υποστηρίζουμε όμως την προσέγγιση σας. Είναι σημαντικότατο να ακολουθήσουμε τη διαδρομή αποκεντρωμένων ευθυνών. Οι πολιτικές και οι κανονισμοί είναι σαν μια μαζεράτη και η τροχή της μαζεράτη είναι, αν αυτό ισχύει σαν μεταφορά, η τροχή της μαζεράτη είναι η, έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Επόμενη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πασίγνωστο ότι η θέρμανση, η αύξηση θερμοκρασία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μία από τι μεγαλύτερε ε, προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Όσον αφορά και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την υγεία και την παγκόσμια οικονομία διάσκεψη του Παρισιού και η συμφωνία που υπεγράφει είναι η αρχή μιας δυναμικής εξελικτικής διαδικασίας που επιτρέψει στην ευρωπαϊκή κοινότητα και τη διεθνή να πετύχει στόχους. Δηλαδή να μειωθεί η αύξηση θερμοκρασίας κάτω από τους δύο βαθμούς Κελσίου και θέλουμε να συμμετέχουν οι μπλεκόμενοι φορείς, να βρούμε μια κοινή απάντηση που θα ανταποκρίνεται στο ύψος των περιστάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο οι περιφέρειες και πόλεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όπως αναφέρθηκε και από τους άλλους συναδέλφους, έχουν ένα ρόλο ουσιαστικό να παίξουν, ούτως ώστε να πετύχουμε τους στόχους, τους κλιματολογικούς σε όλες τις χώρες. Γιατί, διότι μπορούν να επηρεάσουν την κινητικότητα, τις μεταφορές, το σχεδιασμό, τον αστικό, τις κατασκευές, τις οικοδομές, την ενέργεια και τις ε, οικολογικές υποδομές. Χωρίς τη συμμετοχή όλων των φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, πιστεύω ότι οι χώρες δεν θα είναι σε θέση να πετύχουν τους στόχους τους. Η αξιοπιστία των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει τα διάφορα μέρη εξαρτάται επίσης και από την πραγματική συμμετοχή των πόλεων και των περιφερειών, των επιχειρήσεων και των επενδυτών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δώσουν μια ιδιαίτερη προσοχή στη, σύμβαση, ε, στη συνέλευση των δημάρχων για να διατηρηθεί ε, αυτή η προσπάθεια μέχρι το 2030 και μέχρι το 2050 ούτως ώστε να ενθαρρύνουμε αυτή τη δυναμική που υπάρχει σε 6.500 πόλεις και περιφέρειες που έχουν υπογράψει αυτό το σύμφωνο που έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020 και να καταφέρουν ακόμα καλύτερες επιδόσεις. Θεωρώ ότι αυτό το παράδειγμα της συνεργασίας θα μπορούσε να αντιπροσωπεύσει και ένα μοντέλο προς μίμηση από άλλα κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και έτσι θα μπορέσουν να εφαρμοστούν οι αρχές μαζί με άλλες πρωτοβουλίες εθνικό, διεθνές επίπεδο, πρωτοβουλίες που εφαρμόζουν τα δίκτυα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ε, ταυτόχρονα πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να περιθωριοποιήσουμε ποιηθούν οι πόλεις εκείνες που αποφάσισαν να δράσουν για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, αλλά που δεν ανήκουν σε αυτή τη σύμβαση των ε, δημάρχων. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε επίσης ότι οι περιφέρειες και οι πόλεις που συμμετέχουν στην COP21 θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να επενδύσουν. Χρειάζονται σημαντικές καινοτόμε επενδύσεις που θα μπορούν να κατευθυνθούν προς βιώσιμα προγράμματα, κυρίως στον τομέα της ενέργειας, της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων για τις πολύ ε, μικρές κοινότητες. Και θα ήταν χρήσιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να βοηθήσει την εφαρμογή μιας ε, συνεργασίας των διαφόρων τοπικών αρχών, περιφερειακών αρχών και εθνικών αρχών και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο ενιαίο δράσης. Πρόκειται περί των πόλεων και περιφερειών υπέρ του περιβάλλοντος και χρειαζόμαστε όμως εξίσου εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού όσον αφορά τις συνέπειες που έχει η αλλαγή του κλίματος. Όλα τα μέτρα, όλες οι χειρονομίες, ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας στο επίπεδό του για να πετύχει τους βασικούς στόχους αξίζει και πιστεύω ότι η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών πάσης ηλικίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να στέψουμε με επιτυχία την COP21 και να καταπολεμήσουμε πράγματι την αλλαγή του κλίματος. Επόμενος και ο ο κ. Φλακ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ του συντηρητικού του Ηνωμένου Βασιλείου και ευχαριστώ την εισηγήτρια για το επιτελεστέν έργων. Υποστηρίζουμε τις γενικές αρχές του σχεδίου εκθέσεως, όμως κάποια στοιχεία θεωρούμε ότι χρήζουν βελτιώσεων. Δεν υπάρχει κάποια έκπληξη σε αυτό που λέω, φαντάζομαι. Πρέπει να τροποποιηθεί η διατύπωση σε κάποιου σημαντικού τομεί, κυρίω τρει. Πρώτο, όπω ανέφερα και σε πρώτερη ανταλλαγή απόψεων, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να παρακολουθούμε την πραγματική συνεισφορά της πολιτικής συνοχής όσον αφορά την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Το 2016 το ελεκτικό συνέδριο συνεπέρανε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι στόχοι του 20% δαπανών της Ευρωπαϊκής Ενώσης για προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος μέχρι το 2030 ότι δεν θα επιτευχθούν. Χρειάζονται ισχυρότεροι μηχανισμοί εποπτείας. Αυτό πρέπει να έχει προτεραιότητα. Προτείνω σχετική διατύπωση, κυρίως σημειώνοντας την παράγραφο 34 και 35 της νομοδοτήσεως της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε προστιθέμενη αξία που χορηγεί αυτή η έκθεση. Απλώ να δηλώνουμε, παραδείγματο χάρη, ότι είπα θα πρέπει να καταγγελθούν διότι έχουν αποσυρθεί τη Συμφωνία των Παρισίων, όπω γίνεται στην παράγραφο 2, δεν προσθέτει και αξία στην έκθεση που αφορά το ρόλο των πόλεων στην COP21. Με τα χαρά σα άκουσα η να παραδέχεστε σήμερα το πρωί ότι πολλοί μη ομοσπονδιακοί φορείς σε πολιτείες και πόλεις των ΗΠΑ μετά την απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών επινεβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να μειώσουν εκπομπές σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων μέσω πλατφορμών όπως η υπόσχεση δέσμευση της, Αμερικής, της Αμερικής, συγγνώμη, Pledge. Θα πρέπει στην Ευρώπη να δίνουμε την αυτονομία στις περιφέρειες να μπορέσουν να εφαρμόζουν τα δικά τους σχέδια μειώσεως των συνεπειών αλλαγής του κλίματος για να πετύχουν τους φιλόδοξους. Αυτό η σύμβαση των ε, το σύμφωνο των δημάρχων επέτρεψε να ξεπεράσουμε τους στόχους του 20% της Ευρωπαϊκής Ενώσης το 2020. Τρίτον, τελευταίο σημείο. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο θετικοί όσον αφορά το ρόλο της βιομηχανίας. Πολλοί τομεί τη βιομηχανία έχουν δεσμευθεί στην μείωση τη χρήση του άνθρακο και σχετική πολιτική και επενδύουν σε πράσινη τεχνολογία. Όμω, η βιομηχανία επί του παρόντο αναφέρεται μόνο μια φορά στο σχέδιο έκθεση, στην παράγραφο 5. Και θετικά και μετά στα υπόλοιπα σημεία αρνητικά. Η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού τομέα και των περιφερειών έχει οδηγήσει σε πολύτιμε λύσει στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και εντό Ευρωπαϊκή Ενώσεω και σε όλο τον κόσμο. Την περασμένη εβδομάδα η Τέσλα άναψε στην Νότια Αυστραλία τη μεγαλύτερη μπαταρία στον κόσμο. Και αυτή η περιοχή είναι πρωτοπόρος όσον αφορά την αποθήκευση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό χάρη στην Τέσλα. Ε, εξίσου στην Ανατολική Γερμανία, ε, στο Πίτερ Μπορό, στην εγκατάσταση ανάκαμψης, ε, επεξεργαζόμαστε απόβλητα που δεν πάνε στις χωματερές και έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε τα ωφέλη που αποκομίζουμε από την δραστηριοποίηση της βιομηχανίας και θα υποβάλω σχετική τροπολογία. Κατά κλείδι νομίζω ότι έχει γίνει η βασική εργασία, να συμμορφωθούν οι πόλεις με τη Συμφωνία των, ε, των Παρισίων ή με την ομάδα ΣΥΤΕΣ 40 ή με το, το Σύμφωνο των Δημάρχων. Ε, υποστηρίζουμε όμως την έκθεσή σας. Ο κ. Βαν Μιλτεμπερκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο εκ μέρους του κ. Τάκουλα, εκ μέρους του οποίου σας ζητώ συγγνώμη για την απουσία του και θα ήθελα να κάνω ένα-δυο πολύ σύντομα σχόλια, γιατί νομίζω πως ε, έχουμε ήδη ε, υποστηρίξει τις βασικές αρχές αυτής του σχεδίου έκθεση από την πλευρά των φιλελευθέρων της Άντε. Αλλά επιτρέψτε μου να σχολιάσω συγκεκριμένα σημεία. Η παράγραφος 12 καταρχήν. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ρεαλιστική. Μετά από τα όσα ακούσαμε από την πλευρά του Επιτρόπου Ότινα και ο οποίος μας είπε ότι θα πρέπει να αυξηθεί και πάλι ο προπολογισμό ε, της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020. Ίσως αυτό που θα πρέπει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο είναι ότι χρειαζόμαστε την απαραίτητη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων τη κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν δηλαδή πέραν τη περιφερειακή πολιτική και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Ένα δεύτερο ε, σημείο είναι εκείνο ε, του σημείου 14, δηλαδή την υποστήριξη της πολιτικής απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω ε, κατάλληλων προγραμμάτων απασχόλησης. Ναι, αλλά χρειαζόμαστε τέτοιου είδους συγκεκριμένα προγράμματα για όλες αυτές τις προτεραιότητες. Ή μήπως στο πλαίσιο εφαρμογής μιας τέτοιας πολιτικής θα επιτύχουμε ε, περισσότερη απασχόληση. Δηλαδή όταν βλέπουμε στην έκθεση για την πράσινη ενέργεια διαπιστώνουμε ότι πράγματι αυτομάτως υπάρχουν υπάρχει θετικός αντίκτυπος για την απασχόληση. Οπότε χρειαζόμαστε σχέδια απασχόληση ε, τα οποία θα συνοδεύουν την πολιτική απαλλαγή από τι ανθρακούχε εκπομπέ. Ε, Είναι κάτι νομίζω που δεν έχει πολύ θέση ναι. εδώ. Και επίση θα ήθελα μια διευκρίνηση σε σχέση με την παραγράφο 18 όπου αναφέρεστε στην α, εκ των προτέρων αξιολόγηση των κοινων οικονομικών επιπτώσεων των μέτρων. Ε, ναι, προφανώς, το μέτρο προσαρμογή. Προφανώ χρειαζόμαστε μια αξιολόγηση των μέτρων προσαρμογή, αλλά γιατί εκ των προτέρων αξιολόγηση των κοινωνι... κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων αυτών. Ειδικότερα όταν αναφέρεστε στην εστίαση αυτών των μέτρων στην προστασία των πιο ευάλωτων πληστηρισμιακών ομάδων, δηλαδή Ακριβώς επειδή χρειαζόμαστε μετριασμό των επιπτώσεων και χρειαζόμαστε και προσαρμογή, δεν νομίζω πως έχει νόημα να αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, τις οποίες δηλαδή με κάποιο τρόπο θα δώσουμε προτεραιότητα. Γιατί αν το κάνουμε ουσιαστικά δίνουμε την αίσθηση ότι θέλουμε κάποιες κοινωνικές τάξεις οι οποίες είναι πιο ευάλωτες να πρέπει να ε, εποφεληθούν περαιτέρω. Αλλά νομίζω πως αυτές οι, ο μετριασμός των επιπτώσεων και η προσαρμογή του πληθυσμού αφορά το σύνολο του πληθυσμού. Όλοι θα βρεθούμε δηλαδή αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, ο κ. Ε, Ράπε, ο επόμενος αστιώδης συζήτης έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έργο της εδώ πρόκειται για μια σημαντική και απαραίτητη έκθεση, ειδικότερο καθώς ε, ερχόμαστε όλο ένα και πιο κοντά σε μια νέα περίοδο μετά το 2020. Δηλαδή τα όσα έχουμε κάνει σε αυτή την περίοδο από το 2014 έως το 2020 δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε πλέον. Αλλά ε, οι δυνατότητες που θα έχουν οι περιφέρειες και οι πόλεις μετά το 2020 θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για το μέλλον και όπως είπε σωστά η εισηγήτρια σε κάποια σημεία δεν κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία τρέχουν στις διάφορες περιοχές, στις διάφορες περιφέρειες δηλαδή και στις ε, πόλεις και υπάρχουν ευθύνε που έχουν αναλυθεί και δράσει οι οποίε εκτελούνται στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων με βάση τα όσα επιτρέπουν τα ίδια τα κράτη-μέλη, με βάση δηλαδή τι εντολές που δίνουν τα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, στι χώρε τη Βαλτική, Βαλτικής, συγκεκριμένα στη Λιθουανία, οι περιφέρειες είναι αρμόδιε μόνο για το 15% των κονδυλίων χρηματοδότηση και σε πολύ συγκεκριμένου τομεί. και ε, ε, όταν υποχρεωμένε να ακολουθούν πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Άρα για την περίοδο μετά το 2020 θα πρέπει να ε, δώσουμε περισσότερα δικαιώματα σε αυτές τις περιφέρειες, δηλαδή στους πολίτες τελικά, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τουλάχιστον το 50% αυτών των κονδυλίων, προκειμένου να κατευθυνθούν σε σημαντικούς τομείς, για παράδειγμα, όπως η ανακαίνιση των ε, κατοικιών. Για παράδειγμα, ο στόχος ε, που έχει τεθεί είναι ανακαίνιση ε, των όλων των οικειών ε, κατά 3 5%. Τι θα σημαίνει αυτό όμως στην πράξη. Ότι θα χρειαστούμε 60 χρόνια για να ανακαινήσουμε όλα τα ε, όλες τις οικίε. Εμείς όμως έχουμε καταφέρει στην δική μου ε, περιοχή, ε, στο δικό μου δίνο, να προβούμε στην ανακοίνωση όλων των οικειών και επιτυχάνουμε τεράστια εξοικονόμηση ενέργεια. Άρα ενέργειας δεν θα πρέπει να μας ε, απασχολεί μόνο η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Θα πρέπει να μας απασχολεί και η εξοικονόμηση ενέργειας. Ε, δηλαδή το 47% των, ε, ε, της ενέργειας ε, προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και, που καταναλώνουμε εμείς εδώ. Αλλά θεωρώ πως ένα τέτοιο τεράστιο ποσοστό θα μπορούσε να αξιοποιείται αλλού μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας ακριβώς να χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο και υπάρχουν ένα σωρό άλλες σπατάλε τις οποίες προβαίνουμε, για παράδειγμα την απόρριψη ακικών συσκευών, ε, συσκευές τις οποίες πετάμε απλώς και μόνο ε, επειδή κάπου έχει χαλαρώσει μια βίδα. Οπότε θα πρέπει να δοθούν και τα κατάλληλα ερεθίσματα στην βιομηχανία ε, προκειμένου να κατασκευάσουν προϊόντα τα οποία είναι δυνατόν να επισκευάζονται, όχι όπως σήμερα που δεν είναι δυνατή η επισκευή. Άρα λοιπόν ε, θα πρέπει και η κατανάλωση στην οποία προβαίνουμε, στο πλαίσιο ακριβώς της κατανάλωση ενέργειας, να έχει και τα όρια της, να είναι ε, πιο εξορθολογισμένη. Και επίσης σε ό,τι αφορά την, ε, τις αγορές ενέργειας, ήδη αναφέρθηκε ότι οι ΗΠΑ οι οποίες ε, εισάγουν ε, το 50% της ενέργειας τους ε, από άλλες χώρες θα πρέπει να φροντίζουν ότι αυτές οι χώρες θα πληρούν τα ίδια πρότυπα της ασφάλειας τα οποία τηρούμε και εμείς εδώ. Και νομίζω πως υπάρχουν και κάποιες πυρηνικές εγκαταστάσεις ε, οι οποίες ε, κατασκευάζονται αυτή την περίοδο ε, χωρίς όμως να έχει δοθεί, να έχει υπάρξει ένα σχέδιο για την διαχείριση των αποβλήτων, της, αποβλήτων τους. Κατά συνέπεια λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να αποδέχεται στις αγορές της προϊόντα τα οποία ουσιαστικά έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους της και δεν συμμορφώνονται με τις προτεραιότητες στο πλαίσιο της πολιτικής για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Άρα λοιπόν για την περίοδο μετά το 2020 θα πρέπει να μας απασχολήσει ειδικότερα το αν θέλουμε τα κράτη-μέλη να παραμένουν υπεύθυνα για το μεγαλύτερο τμήμα αυτής της πολιτικής ή και οι περιφέρειες θα πρέπει να παίξουν ένα ρόλο. για παράδειγμα στο πλαίσιο της ε, γεωργικής ε, πολιτικής ε, ε, είχαμε διαπιστώσει πόσο καλά λειτουργήσε το σύστημα Leader Plus. Δεν θα μπορούσαμε στο πλαίσιο της ε, ε, πολιτικής εδώ, της περιφερειακής πολιτικής, να έχουμε ένα πρόγραμμα, μια αντίστοιχη προσέγγιση. Δηλαδή, οι περιφέρειες να αποφασίζουν εκείνες ποια είναι τα προγράμματα και πού θα πρέπει να επενδύονται με τον καλύτερο τρόπο τα σχετικά κονδύλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντεμάτο, τώρα και Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα Είμαστε πολύ ευαίσθητοι για αυτό το θέμα που αναφέρει η έκθεση κυρίως για την αλλαγή του κλίματος. Εξαιτία τη αλλαγή του κλίματο, οι ευρωπαϊκέ περιφέρειες είναι υποχρεωμένε να αντιμετωπίσουν μετεωρολογικά γεγονότα όπω η ξηρασία, οι θύλε, οι πλημμύρε, που με αυξανόμενη ένταση και συχνότητα εμφανίζονται. από Το 1980 μέχρι το 2013 υπολογίζονται ζημιέ οικονομικέ περίπου ύψου 400 δισεκατομμυρίων και μιλούμε μόνο για την πτυχή την οικονομική και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος μας ζητά να μελετήσουμε στατηγικές πολιτικές και μέτρα προσαρμογής που είναι καλύτερα ε, και πιο ευέλικτα. Να θυμηθούμε ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, το 20% του ευρωπαϊκού προπολογισμού για την περίοδο 2014-2020, θα έπρεπε να δαπανηθεί για δράσεις που αφορούν το κλίμα. Όμω, ε, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του του 2016 μας λέει ότι υπάρχει κίνδυνος να μην καταφέρουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Μετά υπάρχει και μια άλλη πτυχή. Λοιπόν, η πτυχή των ζημιών που σχετίζονται με τη βιπικιλότητα ε, πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη και την ανθρώπινη υγεία ε, που δεν αναγνωρίζεται πολύ συχνά και ε, υπάρχει μια άρνηση ανά αυτών των συνεπειών. Ήδη με τρόπο έχουν, έχουμε πρόημους θανάτους και ασθένειες από, τις, από αυτά τα φαινόμενα. Και η ατμόσφαιρα έχει γίνει πιο ε, θανατηφόρα από το 2015 και έχει οδηγήσει σε χιλιάδες θανάτους. Έχουμε πλημμύρες, ε, παράκτιες, ποτάμιες ε, και έχουν ε, σκοτωθεί και έχουν πληγεί πολλοί άνθρωποι. Αυτά επηρεάζουν αρνητικά ε, έχουν τραυματισμούς, μολύνσεις, εκθέσεις σε χημικούς κινδύνους και στρες. Δημιουργούνται αυτοί οι κίνδυνοι για την υγεία και διακόπτονται υπηρεσίες όπως στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης ε, για μακρές περιόδους. Λοιπόν, κάτι αναφέρεται στην παράγραφο 9 και 10 σχετικά με αυτό, όμως εμείς θα υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες για να συμβάλλουμε στο έργο που έχει κάνει η συγκήτρια. Εκτιμούμε και πολύ το χρειάζεται επί των πόλεων γνωρίζουμε ότι είναι σημαντική η αντοχή των πόλεων των ευρωπαϊκών αντί του κλίματος που φιλοξενούν τα τέταρτα του πληθυσμού και είδαμε τα φοβερά γεγονότα στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα, στην Γαλλία την, ε, και την Ιταλία, στην Νότια Γαλλία και έδειξαν ότι τελικά έχει μειωθεί η απόσταση μεταξύ, λόγω της επεκτάσεως των πόλεων έχει μειωθεί η απόσταση μεταξύ των ε, ε, δασικών περιοχών και των πόλεων. Πρέπει να αυξήσουμε και την αύξηση του, του προπολογισμού που αφιερώνεται σε αυτό το πρόβλημα μέσω της πολιτικής συνοχής για να αντισταχθούμε ε, στην αλλαγή του κλίματος με συγκεκριμένους στόχους. Χρειαζόμαστε καλύτερα κίνητρα για ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την πρόληψη ε, των αλλαγών λόγω του κλίματος και θα πρέπει να προτείνουμε και μια αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης μέσω της εκθέσεως. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ε, υπάρχουν... Α, η κυρία Κρέλ, κυρία Κρέλ; Ναι, κυρία Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο πράγματι γιατί θα ήθελα να πω δύο πράγματα κι εγώ. Ε, ε υποστηρίζω πλήρως ε, στόχους ε, που έχει θέσει η συγχύτρια. Απλώς θα ήθελα να κάνω τρία σχόλια. Στο σημείο 5, όπου κάνετε μια γενική περιγραφή, ε, αναφέρατε κάτι το οποίο ίσως ε, να μην κατάλαβα καλύτερα και με τη διερμηνία. Εδώ στα γερμανικά τι βλέπω. Ε, να λέτε, εκφράζει τη λύπη του για τη σοβαρή ανευθυνότητα των κλάδων τη βιομηχανία, τη επικοινωνία και τη πολιτική που συνεχίζουν να αρνούνται τα αποδεικτικά στοιχεία τη αλλαγή του κλίματο. Τι σημαίνει αυτό στα γερμανικά. Δηλαδή, όλοι οι πολιτική, όλα τα μέσα ενημέρωσης ουσιαστικά ψεύδονται σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Ε, εκείνο που λοιπόν που θα πρέπει να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον κλάδο, τη, τη βιομηχανία δηλαδή, προκειμένου να αξιοποιεί τέτοιες τεχνολογίες, για παράδειγμα, οι οποίες εξοικονομούν τις πρώτες ύλες, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ε, δηλαδή έτσι απλά αυτή η έκφραση δεν ισχύει. Και οι ίδιοι είμαστε πολιτικοί. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι ενδέχεται να αρνούνται αυτή την κλιματική αλλαγή, αλλά ε, και εδώ έχουμε και το παράδειγμα του Προέδρου Τραμπ, αλλά σίγουρα δεν είμαστε όλοι. Οπότε θα πρέπει να διατυπωθεί αυτό το σημείο διαφορετικά, σε διαφορετική περίπτωση ε, δίνει λανθασμένη εντύπωση. Επίσης, με αυτό το ψήφισμα δεν νομίζω πως θα πρέπει να προδικάσουμε το ύψος των κονδυλίων ε, που θέλουμε να επενδύσουμε στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτή τη στιγμή το 20% των συνόλων των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής έχουν κατευθυνθεί προς αυτούς τους στόχους και είναι σωστό αυτό, αλλά δεν νομίζω πως θα έπρεπε από τώρα να πούμε ότι το λόγο ποσοστό θα πρέπει να αυξηθεί. Θα πρέπει να δούμε ε, ποια θα είναι η πρόταση που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του επόμενου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου και μετά να αποφασίσουμε. Αλλά σίγουρα συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τι πόλει έτσι ώστε να μπορούν οι ίδιε να αποφασίζουν ε, ε ποιε θα είναι οι δαπάνε ε, στο πλαίσιο τη επιδίωξη αυτών των στόχων. Δηλαδή έτσι ώστε να μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα στο πλαίσιο τη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με αυτόν τον τρόπο θα ήταν δυνατό να εργαστούν εντατικότερα για την καταπολέμηση ε, τη κλιματική αλλαγή, είτε πρόκειται στον κατασκευαστικό τομέα, δηλαδή κατασκευή κατοικιών, είτε πρόκειται στον τομέα των μεταφορών εντό των πόλεων και ούτω ε, καθεξή. Νομίζω λοιπόν πω με αυτέ τι διορθώσει θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλου ε, συμμετέχοντε. Θα ήθελα να δώσω λόγο το λόγο στην κυρία Μαλινόφσκα από την Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και αγαπητά μέλη για τη συζήτηση. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί χρειάζεται κινητοποίηση και δράση για αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Τώρα επιστρέψαμε από τη Βόνη, από την διάσκεψη τα μέσα Νοεμβρίου και θα γίνει και μια συνάντηση την επόμενη εβδομάδα στο Παρίσι. Οι τοπικές αρχές και οι περιφερειακές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Στη διάσκεψη η συμμετοχή των δημάρχων και των τοπικών αρχών οδήγησε ε, στη συμμετοχή 300 πολιτικών αρχηγών και χιλιάδων συμμετεχόντων από 60 χώρες, συμπεριλαμβάνοντας και τα μικρά νησιά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή των Περιφερειών που ε, διοργάνωσε αυτή την ε, συμμετοχή των δημάρχων, καθώς και την διατλαντική συνεργασία, την διευκόλυνση χρηματοδότησης και την ε, πολιτική ε, ηγεσία σε αυτό το τομέα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ πόλεων, εθνικών κυβερνήσεων και περιφερειών μέσα στα πλαίσια καινοτόμων λύσεων και του κρίσιμου ρόλου των ε, βιομηχανιών, καθώς ε, και τη συνέργεια δημόσιου ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις στην ε, ε, Βόνη μιλήσαμε για ένα διάλογο τύπου Ταλανόα όπου οι μεγάλες και μικρές πόλεις ε, θα συνδράμουν για να δούμε πόσο κοντά βρισκόμαστε σε αυτές τις δεσμεύσεις και για να επιταχυνθεί η διαδικασία των Παρισίων ως προς το προσχέδιο γνωμοδότησης που συζήτηση σήμερα το δεχόμαστε ε, φυσικά είναι απόλυτα ευπρόσδεκτο μέσα στα πλαίσια των απότερων στόχων για καθαρή ενέργεια, για προτάσεις περί καθαρής ενέργειας αλλά θα πρέπει να τονίσουμε τον ρόλο των ε, εθνικών φορέων. Επίσης, ε, αναζητούμε την άποψη πολλών ε, πόλεων της Ευρώπης για δράση υπέρ του κλίματος και κατά των αλλαγών. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχε μία μεγάλη συνδρομή στη Βόνη από τις πόλεις και φυσικά υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ε, προώθησης της ε, ποιότητας εργασίας και της υγείας. Από πλευράς πολιετούς θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνδράμουμε περισσότερο χρηματοοικονομικά, διότι οι δεσμεύσει των Παρισίων ε, είναι μαζικές και φυσικά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτή την δημοσιονομική σύνδρομη όπως προτείναμε στο Παρίσι. Επίσης ε, υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα χρήματα για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και διαχείριση κινδύνων, ένα ως προς ε, τη θεματική αυτή προσπάθεια και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να βοηθήσουμε πόλεις και περιφέρειες για να υπάρχει μεγαλύτερη ε, ενσυνειδητότητα για προσαρμογή και απάλυνση των ε, επιπτώσεων και σε επίπεδο δημάρχων από τον παρελθόντα σε Σεπτέμβριο είδαμε ότι εργαζόμαστε συστηματικά για, τις, ε, την υποσαχάρια περιοχή καθώς και για την Αμερική και την Ινδία. Την προηγούμενη εβδομάδα ε, έχουμε ήδη προωθήσει το σχέδιο Ούρπης ε, για την συνδρομή πόλεων με την βοήθεια και της ΕΤΕΠ για να μπορέσουμε να προωθήσουμε συγκεκριμένα σχέδια. Γιατί υπάρχουν τα χρήματα, όμως δεν προσδένονται σε συγκεκριμένα σχέδια. Και όπως προαναφέρθηκε εδώ, η συνδιάσκεψη των δημάρχων συνδράμει στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Μιλάμε για ένα 23% μείωση και ε, έχουμε φτάσει ήδη στο 27% των ε, δεσμεύσεων. Χιλιάδες πόλεις ε, συνδράμουν και θεωρώ ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις κατέχουν ηγετικό ρόλο για να φτάσουμε σε ένα μεγάλο εγχείρημα επιτυχίας ανά τον κόσμο. Η κυρία Βαλίνα έχει το λόγο τώρα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για... και σε εσά σε όλους και στην εκπρόσωπο της Επιτροπής. Εγώ προέρχομαι από μια περιφέρεια όπου τα ανθρακοριχεία ήταν η βασική πηγή εσόδων της περιοχής και φυσικά και οι συναφείς βιομηχανίες, όταν υπήρχαν αυτές οι βιομηχανίες. Και όπως ξέρετε, εκεί ε, συγκεντρώνονταν οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Φυσικά δεν μπορούμε να ε, ζήσουμε χωρίς τη βιομηχανία, αλλά θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις ε, ε, περιβαλλοντικές προσταγές. Γιατί εγώ ήμουν δήμαρχος για εννέα χρόνια σε αυτή την περιφέρεια και χρειάστηκε να ανασύρουμε βαρέα ε, μέταλλα πολύ κοντά στις, στην παραλία όπου έκαναν μπάνιο οι άνθρωποι και όπου δρούσε αυτή η μεγάλη βιομηχανική μονάδα. Όμως ε, η βιομηχανία πρέπει να ε, μπορέσει να δεσμευτεί και να υπάρχει και δέσμευση ως προς την απομάκρυνση από τη χρήση του άνθρακα, γιατί εμείς είχαμε 50.000 ανθρακορίχους τότε και τώρα έχουμε 800 μόνο ανθρακοριχούς. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει απερίμωση αυτών των περιοχών και μετανάστευση. Ναι, φυσικά θα πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους μία εναλλακτική όταν ε, τους αποστερούμε την εργασία. Γι' αυτό η απομάκρυνση από τον ανθρακά θα πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους να έχουν ε, ένα εισόδημα και μία αξιοπρεπή ζωή. Γιατί έχασαν την εργασία τους και έχει πολύ μεγάλη σημασία η συνδρομή των δημαρχείων, των τοπικών αρχών. Στην Ισπανία έχει γίνει μία μεταρρύθμιση για την αυτονομία των περιφερειών. Εγώ εργάζομαι στην Επιτροπή Αναφορών και εκεί βλέπουμε συνεχώς αναφορές για προστατευόμενες περιοχές όπου υπάρχουν ε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ε, συγκεκριμένη έλλειψη προγραμματισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τις περιφέρειες και τις ε, τοπικές αρχές. Δεν μπορούμε όλοι να ε, βασιζόμαστε σε ένα γραφείο ή στο, στο συγκεντρωτισμό ενός ε, κράτους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις υποδείξεις και αναμένω προτάσεις τροπολογιών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το μόνο που πρέπει να πω στο τέλος της συζήτησης είναι ότι η προθεσμία τροπολογιών είναι το μεσημέρι της Τετάρτης 13ης Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και τώρα μεταβαίνουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης για να μην κάνω λάθος αυτή τη φορά, η ανταγωνιστικότητα στις περιοχές που παρουσιάζουν ε, αναπτυξιακή καθυστέρηση. Η κυρία Τζουφρίντα είναι η, η συγγήτρια και σήμερα θα συζητήσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης. Η κυρία Τζουφρίντα έχει το λόγο ή θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά πιστεύω ότι η συζήτηση από αυτές τις περιοχές αυτές ε, που έχουν καθυστερήσει είναι κάτι πολύ σημαντικό για την πολιτική συνοχή. Γι' αυτό Δοθέντω ότι η έκθεση είναι έτοιμη σχεδόν, εγώ είμαι έτοιμη να ακούσω τις συστάσεις των ε, συναδέλφων. Είναι οι πιο αδύναμες περιοχές της Ευρώπης αυτές που έχουν μείνει πίσω, που εξορισμού είναι οι πρώτοι αποδέκτες της πολιτικής συνοχής και οι περιοχές τις οποίες πρέπει πάντα να υποστηρίζουμε και να τι έχουμε υπόψη. Χρειάζεται και ευρωπαϊκή υποστήριξη. Είναι χρήσιμο που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία που εξετάζει τους παράγοντες, περιορίζουν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη των περιοχών με αναπτυξιακή στέρηση, δηλαδή περιοχές με χαμηλό εισόδημα και με χαμηλή ανάπτυξη. Αυτές είναι οι διακρίσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, πάνω σε αυτές τις διακρίσεις κινείται η έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοπτικά στη μελέτη εντοπίζει 47 περιοχές με αναπτυξιακή στέρηση, τις υποδιαιρεί με χαμηλή ανάπτυξη, τις περιοχές που έχουν ένα ΕΠ που πλησιάζει το μέσο όρο της Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όσον αφορά την οικονομική, έχουν οικονομική ανάπτυξη ε, που είναι σε πολύ χαμηλου ρυθμού. Παράδειγμα, έχουμε διάφορες περιοχές χωρών όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Ελλάδα και όπως είναι η Πορτογαλία. Δεύτερη διαφοροποίηση αφορά τις περιοχές με χαμηλό εισόδημα. Περιοχές με ένα ΕΠ που είναι ακόμα πολύ χαμηλό, αλλά που έχουν μία τάση αναπτυξιακή ε, αξιοσημείωτη που ξεκινούσαν από μία ιστέρηση πολύ μεγαλύτερη από αυτές που προανέφερα, αλλά όπου η πολιτική συνοχής λειτουργεί αποτελεσματικά, όπου καταγράφονται πολύ καλά αποτελέσματα χάρη στη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων. Και για να δώσω κάποια παραδείγματα, εδώ μιλάμε για περιοχές που ανήκουν σε χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ρουμανία. Αυτό που θα ήθελα να πω καταρχάς είναι ότι πάνω απ' όλα αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να ισχύει για λόγους μελέτης και στατιστικών στοιχείων, όμως δεν είναι κάτι που προέρχεται τους κανονισμούς. Και πιστεύω ότι το να κάνουμε τέτοιου είδους ταξινομήσεις είναι κάτι που θα οδηγούσε σε μια υπερβολικά και πιθανότατα μια αποτελεσματικ... ένα... μια αποτελεσματικό κατακαιρματισμό. Πρέπει να σχετίζουμε και με ε, περιόδους αναφοράς που ταιριάζουν και με τις περιόδους και τρόπους χρηματοδοτήσεως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοιτά ποιε είναι οι συνέπειε, ποια είναι τα αποτελέσματα τη πολιτική συνοχή σε αυτές τις περιοχές και τι συσχετεί τα αποτελέσματα την οικονομική ε, κατάσταση τη χώρα στην οποία ανήκουν οι περιοχέ, λέγοντα ότι το μεγάλο δημόσιο χρέο ε, περιορίζει τις δυνατότητες ελιγμών ε, του, στον προϋπολογισμό και την χρήση των ε, ταμείων. Όμως αυτές τις διαφοροποίησεις και η προσεγγίση Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας οδηγεί στον κίνδυνο να απομακρυνθούμε από τους πραγματικούς στόχους και την έννοια των ε, πολιτικών συνοχής. Και πιστεύω ότι είναι η στιγμή, το αναφέραμε αυτό και στη συζήτηση που προηγήθηκε, ε, να διεκδικήσουμε τον πολιτικό μας ρόλο, που είναι διαφορετικός προφανώς από αυτόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προτείνουμε κάποιες πολιτικές φύσεως λύσεις. Ενετόπισα τρία σημεία διαφορετικά στην έκθεση για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ πολιτικής οικονομίας, μεταξύ συνοχής και οικονομικού governance. Μια ισορροπία που μπορεί να υπονομευθεί ήδη στο εγγύς μέλλον λόγω των αλλαγών που ζούμε. Με μια πολιτική συνοχής που θα ελέγχεται από την πολιτική οικονομική έτσι έχει κατάσταση. Στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναφέρει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει την τοπική αυτοδιοίκηση όσον αφορά τις επενδύσεις. Και αναφέρομαι στις παραμέτρους όσον αφορά το έλλειμμα και τα όρια του προπολογισμού. Πιστεύω ότι αν θέσουμε τροχοπέδι στις επενδύσεις ε, ε, ε, τα περισσότερα όρια τίθεται από τον πέρα από την πολιτική συνοχής δημιουργεί απασχόληση και ανάπτυξη πολιτικής συνοχής. Αλλά το πρόβλημα είναι η συγχρηματοδότηση που διέπεται και από το Σύμφωνο Σταθερότητας. Και επιμένουμε από αυτού. Μετά πρέπει να δούμε το μηχανισμό της αιρεσιμότητας μακροοικονομικής. Πρέπει να διευθυνθεί να μην κινδυνεύσουν οι επενδύσεις, όπως το είδαμε σε άλλες περιπτώσεις, σε περιοχές εκείνες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες διαθωτικές δυσκολίες. Πρέπει να σεβαστούμε τις, μακροοικονομικέ μακροοικονομικές παραμέτρους και υπάρχουν και άλλες αιρεσιμότητες στην περίπτωση της ε, συνοχής, όπως και άλλες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα πρέπει να επικεντρώνονται οι αιρεσιμότητες στο ε, σεβασμό των θεμελιωδών αξιών και στη συμβίωση που είναι βασικό μας πιστεύω. Λοιπόν, η ρεσιμότητα η μακροοικονομική θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σαν μια παράμετρος για την ενεργοποίηση μέτρων συνοχής με μια οπτική θετική και επικοδομητική δηλαδή για να δοθούν κίνητρα και να τονωθούν οι μεταρρυθμίσεις. Τρίτο και τελικό σημείο, ε, το οποίο αφορά ε, το σημείο που θέλει καλύτερη σχέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ πολιτικής συνοχής και μεταξύ συγκεκριμένων ε, συστάσεων για τις χώρες στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Δεν μας λέει πώς όμως θα γίνει αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι οι συστάσεις δεν θα πρέπει να είναι ένας δεσμός, αλλά ένα κίνητρο που θα στηρίζει τις περιφέρειες. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ένας θετικός κύκλος ε, αένος συνεργασίας μέσω κινήτρων για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που εντοπίζονται από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά. Θα πρέπει, όπως έλεγα, να βρούμε ε, νέα ισορροπία μεταξύ εξουσιών. Από από τον ορισμό τη πολιτική συνοχή στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να ξεκινήσουμε. Θα δούμε ποιε είναι ευρωπαϊκέ ε, οικονομικές πολιτικές και εκεί πρέπει να παίξουν και θεμελιώδη ρόλο και τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να θετήσουν εθνικές στατικές τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη των περιφερειών με οικονομική στέρηση. Μια προσέγγιση που θα συμμερίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου πρέπει να υπογραμμίσω και το αναφέρει, αναφέρει τη χώρα μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το υποστηρίζω και εγώ. Παίρνει σαν παράδειγμα την Ιταλία και τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν στην Ιταλία πρόσφατα με, το σύμφωνο για τον Νότο, για τις μειονεκτούσες περιοχές που βρίσκονται στον Νότο κυρίως, δημιουργία της υπηρεσίας για τη συνοχή είναι ένας φορέας που συνοδεύει τις ε, περιφέρειες όσον αφορά τις δαπάνες και στη σωστή χρήση των πόρων και που εφαρμόζει συνεχή έλεγχο. Λοιπόν, βασική αδυναμία των υστερούντων περιοχών ε, οφείλεται στη διακυβέρνηση και στη διοικητική καθυστέρηση. Και τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να παρέμβουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ξέρω πολύ καλά ότι πρόκειται περί επιμάχων ζητημάτων. Επ' αυτών πολύ συχνά δεν έχουμε βρει ε, μια ενιαία θέση εδώ στην Επιτροπή. Αντιθέτως ε, πολύ συχνά έχουμε συγκρουστεί. Εγώ ελπίζω σε αυτή την περίπτωση πραγματικά να υπάρξει μια ενότητα προθέσεων διότι στις συζητήσεις μας των τελευταίων μηνών είδαμε ε, πως η ενότητα και συμπαγής κίνηση είναι κάτι πολύ σημαντικό τόσο ώστε να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους μέσω της πολιτικής συνοχής. Περιμένω να ακούσω τις απόψεις σας και να δω τις συνεισφορές σας, αλλά κρίνοντας πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή όλος ιδιαίτερος η Επιτροπή μας έχει ιδιαίτερη ευθύνη έναντι αυτών των περιοχών ε, όπως και εκείνες έχουν έναντι της Ευρώπης χωρίς να έχουμε θετική ε, προσέγγιση, θα βοηθήσουμε τις περιοχές να αναπτυχθούν και να βοηθήσουμε και την Ευρώπη να κινηθεί προς μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Ευχαριστώ την προσοχή σας. Περιμένω να ακούσω παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθούμε το άρθρο 54. Είμαστε μαζί με την, περιοχή, με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ο κύριος Τσίλα, η κυρία Τσίλα είναι υπεύθυνη και μετά θα δώσω τους ε, σκέους μετά της δικής μας Επιτροπής το λόγο, αφού ακούσουμε την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται η πιο πλούσια περιφέρεια του κόσμου, όμως υπάρχουν μεγάλες ε, αποκλίσεις ενδοκινοτικά εξαιτίας ε, ε, διαφορετικών επιπέδων ε, εισοδήματος. Περίπου 407 περιφέρειες ε, δυστυχώς έχουν χαμηλό εισόδημα ε, ή χαμηλή ανάπτυξη. Η πρώτη ομάδα βρίσκεται στο νότο της Ευρώπης, ενώ η δεύτερη στην Ανατολική Ευρώπη. Θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της γεωργίας και πώς η γεωργία μπορεί να μας δώσει προστιθέμενη αξία για την αντιμετώπιση των μεγάλων αποκλίσεων. Καθίσταται σαφές ότι σε πολλές περιφέρειες η γεωργία είναι βασικός, ε, βασική πηγή εισοδήματο μέσα στα πλαίσια του πυλώνα της γεωργικής πολιτικής και της περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει μεγάλη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη των ε, γεωργικών περιφερειών που έχουν μείνει πίσω και φυσικά χρειάζεται και η συναφής χρηματοδότηση. Η γεωργία μπορεί να δώσει θέσεις εργασίας και σε περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος, αλλά και σε περιφέρειες με χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και αύξηση εισοδήματος, συνεισφέροντας ε, στην καταπολέμηση της απερίμωσης αυτών των περιοχών. Επίσης, ε, έχουν μεγάλη σημασία τα κονδύλια ε, για την ε, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και φυσικά μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων. Θεωρώ σημαντική και ευπρόσδεκτη τη συνεισφορά των τοπικών φορέων για την εκπόνηση τοπικών στρατηγικών και ανάπτυξη δικτύων, αξιολόγησης ε, και έγκρισης προγραμμάτων ε, leader. Θεωρώ θα, ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί το ευρυζωνικό ε, και στις αγροτικές περιοχές καθώς και η συμμετοχή μίας, ε, ε, ενός εργατικού δυναμικού που να έχει τα κατάλληλα προσόντα. Η ψηφιακή συμμετοχή είναι ύψης της σημασίας και στον τομέα της έρευνας και της ε, Ευρωπαϊκής Εταιρικότητας για την καινοτομία για να προωθήσουμε την γεωργική ανάπτυξη καθώς και τις επιχειρήσεις και τέλος θα πρέπει να προωθήσουμε την ε, οικονομική ανάπτυξη αυτών των περιφερειών που παρουσιάζουν πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ο κύριος Ρούας τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι εδώ και τρεις μήνες μιλήσαμε για πρώτη φορά για αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ανάπτυξη των περιφερειών, ιδιαίτερα αυτών που παρουσιάζουν μεγάλη αναπτυξιακή καθυστέρηση. Νομίζω ότι οι θέσεις αυτής της έκθεσης αποτελούν μία πολύ καλή βάση εργασίας, ιδιαίτερα για τις περιφέρειες που βρίσκονται σε ύφεση. Και φυσικά δεν μπορούμε να αφήσουμε κατά μέρος τις συνθήκες ε, προώθησης του επιχειρήν πάντα υπάρχουν περιθώρια για να ε, διευρύνουμε την συμμετοχή των επιχειρήσεων και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά θα υποβάλω και σχετικές τροπολογίες. Προσπαθούμε να συνδράμουμε σε αυτή την πτυχή του ζητήματος που προανέφερα μέσα στα πλαίσια της πρώτης ανταλλαγής απόψεων. Μιλάμε για την ε, ε, διακυβερνητική συμμετοχή, για την εκπόνηση επιμέρους στρατηγικών για κάθε περιφέρεια, έτσι ώστε και η Eurostat Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσουν να μας δώσουν δεδομένα τα οποία να είναι αξιόπιστα. Οπωσδήποτε όλα αυτά ε, έχουν ήδη εκπληρωθεί εν μέρη από την Κομισιόν. Θα συζητηθούν και οι συναφείς τροπολογίες και από τους σκιώδεις. Θα ήθελα να μιλήσω για την μακροοικονομική αιρεσιμότητα και θα υποβάλω ορισμένες τροπολογίες ως σκιώδεις από το ΕΛΚ. Η έκθεση βέβαια αυτή δεν αφορά την μακροοικονομική αιρεσιμότητα, αλλά την πολιτική συνοχής. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τις ε, περιοχές που βρίσκονται σε ύφεση ιδιαίτερα για να μπορέσουμε να τις συνδράμουμε κατάλληλα. Πάντα γίνονται ζωηρές ε, συζητήσεις επί του θέματος, αλλά πολλές φορές ε, δεν συνδράμουμε επαρκώς θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει, να υπάρξει μια χρηστή ε, οικονομική διαχείριση και η εφαρμογή αυτών των μέτρων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη της, ε, την οικονομικοκοινωνική πραγματικότητα της κάθε περιφέρειας καθώς ε, και τη συμμετοχή των περιφερειακών ταμείων για τις ε, ΜΜΕ για να προσπαθήσουμε να δώσουμε όθεση στην ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες. Πέρσι ήμουν από τους πρώτους που μίλησαν για την εφαρμογή αυτού του πλαισίου στην Ισπανία και Πορτογαλία. Πρόκειται για, επρόκειτο για ανεπαρκή μέτρα γι' αυτό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ερεσιμότητες εξ άντε για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη χρήση των ε, διαρθρωτικών ταμείων όπως έχουν καταδείξει και οι συναφείς έρευνες. Θα πρέπει λοιπόν να φτάσουμε σε μια κοινή θέση και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ορίσει νέους κανόνες για το επόμενο πολιετές. Όπως ήδη έχω προαναφέρει, θα πρέπει να ε, εξορθολογήσουμε τα μέτρα που προβάλλονται από το άρθρο 23 του πολιετούς ε, δημοσιονομικού και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε περίπτωση αναστολής πληρωμών από τα διαρθρωτικά ταμεία. Και φυσικά ε, η καλύτερη λύση είναι στην χρυσή τομή που μπορούμε να βρούμε και στην οποία μπορούμε να φτάσουμε για να μπορέσουμε να συγκλίνουμε σε μία οριστική θέση. Γιατί αυτό είναι, αυτή είναι και η θέληση των πολιτών που μας εξέλεξαν. Θα υποβάλουμε συναφείς τροπολογίες και πιστεύω ότι θα φτάσουμε και σε τροπολογίες συμβασμού, εάν το επιθυμεί η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σίτσου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια πρωτοβουλία προκειμένου να υποστηριχθούν ε, στην προσπάθεια τους ε, να ε, ανακτήσουν το χαμένο έδαφος στις περιοχές. περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή προσπαθούμε να δώσουμε ελπίδα σε αυτές τις περιοχές και να παράσχουμε συστάσεις και υποστήριξη έτσι ώστε να απελευθερώσουν το αναπτυξιακό τους δυναμικό. Οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές με αυτόν τον τρόπο ε, θα μπορέσουν να αναγνωρίσουν και να ανταποκριθούν καλύτερα στις πιο σημαντικές ανάγκες τους έτσι ώστε το, οι επενδύσεις επιτόπι να έχουν ε, ακόμα μεγαλύτερο αντίκτυπο. Η Επιτροπή ε, συνεργάζεται με τις αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η πρακτική εμπειρογνωμοσύνη για, την, ε, για να υπεκεραστούν τα εμπόδια και να υπάρξει περισσότερη επένδυση στις ε, υποδομές και στην καινοτομία. Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες ε, που υποστηρίζω είναι ε, το υψηλότερο επίπεδο εμπλοκής των ε, τοπικών φορέων, των ακαδημαϊκών οργανώσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων, αλλά και των κυβερνητικών αρχών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η Ρουμανία και η Πολωνία ανέλαβαν τον ηγετικό ρόλο σε αυτή την πρωτοβουλία με αντίστοιχες περιοχές στα βόρεια-ανατολικά και στα βόρεια-δυτικά. Ε, στο Πιετοκύρσκι και στο Πόρτ Καρπάσκι. Ε, και ε, αυτό το μοντέλο συνεργασίας ε, στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτού του project ε, που συμπεριλαμβάνει δηλαδή τη συμμετοχή και των τοπικών φορέων θα μεταφερθεί και σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Ελπίζω λοιπόν πως θα ενθαρρυνθούν οι υπόλοιπε περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσουν αυτή την πρωτοβουλία. Οι κύριες ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιοχές με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης είναι η αναγνώριση και η χάραξη στρατηγικών που θα τους επιτρέψουν να ξεφύγουν από ένα διέξοδο στο οποίο βρίσκονται εδώ και δεκαετίες. Ε, η κύρια πρόκληση αυτών των περιοχών είναι η βιωσιμότητα ε, της ε, αναπτυξιακής τους άγουσας και η δυνατότητά τους να ξεκινήσουν μια νέα αναπτυξιακή πορεία η οποία ακριβώς θα τους επιτρέψει μακροπρόθεσμα να αναπτυχθούν. Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να σταθεροποιήσουν την οικονομική τους ανάπτυξη έτσι ώστε να ε, έρθουν και πάλι σε πορεία σύγκληση με τις πιο ευημερούσε περιοχέ τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Βαμίλτεμπουργκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κατά τη δική μου άποψη, η ε, πρόταση αυτή έκθεση δεν είναι ισορροπημένη. Γιατί εδώ αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι ε, να, ε, ακριβώς να βρούμε μια ισορροπία σε ό,τι αφορά τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα αφενός και την πολιτική συνοχή αφετέρου. Ε, η συγκέντρια μας λέει ότι ουσιαστικά όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι λιγότερο ε, ανεπτυγμένες περιοχές οφείλονται ουσιαστικά σε αυτήν την έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στις μακροοικονομικές αιρεσιμότητες αφενός και την πολιτική συνοχή αφετέρου. Δεν αναφέρει δηλαδή τίποτα ως προς την άμεση ανάγκη επενδύσεων από την πλευρά τον ίδιο τον, ε, ή τις ίδιες τις ε, λιγότερο αναπτυγμένε, τι θερούσες ε, περιοχέ. Οπότε νομίζω πραγματικά πως αυτή η πρόταση έκθεση ουσιαστικά ακολουθεί μια πολιτική στοθοκαμιλισμού. Δηλαδή ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας, δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, να αναγνωρίσουμε τα προβλήματα της κυβέρνησης σε αυτές τις περιοχές. Δεν γίνεται λόγος για παράδειγμα τη διαφθορά, δεν γίνεται λόγος για επενδύσεις στην υποδομή, δεν γίνεται λόγος ε, για, την, ε, ε, για μια προσπάθεια αναθεώρησης, αναδιαμόρφωσης της πολιτικής απασχόλησης. Ε, το έγγραφο εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται σε όλα αυτά τα σημεία και με υποδειγματικό τρόπο, αλλά η πρόταση έκθεση τη συγκέντρωση δεν το κάνει. Ε, οι πιο αδύναμε περιοχέ, ειδικότερα εκείνε με χαμηλού ρυθμού ανάπτυξη, ε, έχουν συχνά προβλήματα δημοσιονομικού χαρακτήρα σε σχέση με τον προπολογισμό του γιατί ακριβώ είναι υπερχρεωμένε. Και ε, με αποτέλεσμα όλες, όλα τα φορολογικά έσοδα να κατευθύνονται για την εξυπηρέτηση των χρεών τους. Για το οπότε, για τα χρεολύσια, συγγνώμη, οπότε ε, δεν τους απομένουν κονδύλια τα οποία μπορούν να κατευθυνθούν σε επενδύσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε εμείς τώρα ότι θα πρέπει να υπάρξουν υψηλότερα, κρατικέ ε, υψηλότερες κρατικές δαπάνες για αυτές τις ε, περιοχές. Όχι και στο έγγραφο εργασίας της η Επιτροπή αναφέρει έναν έξυπνο τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί υψηλότερο δυνατό ανάπτυξη, ειδικότερα του ιδιωτικού τομέα, ο οποίο θα είναι και πολύ λιγότερο, θα εξαρτάται πολύ λιγότερο από τι δημόσιε επενδύσει και κατά συνέπεια θα είναι και πολύ λιγότερο ευάλωτο σε περίπτωση ε, ε, οικονομική ύφεση. Υπάρχουν λοιπόν μία σειρά από διαφορετικέ λύσει που προτείνονται και στο έγγραφο εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τι οποίε δεν θίγει η εισηγήτρια. Δηλαδή, πώ μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε την αγορά εργασία, πώ μπορούμε να προβούμε σε επενδύσει στην υποδομή. Έχουμε δει πώ έχουν λειτουργήσει τέτοιε πολιτικέ. Για παράδειγμα, στις, ό,τι αφορά την κατάσταση των ανθρώπων στην Ρουμανία. Στη Ρουμανία είναι απολύτω απαραίτητε τέτοιου είδου επενδύσει στι υποδομέ. Και αυτό σχετίζεται και με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. και αυτό το ζήτημα αναφέρεται στο έγγραφο εργασία της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Αναφέρεται επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στις ε, πόλεις οι οποίες αποτελούν την, ε, την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και τι γύρω περιοχέ τους. Τίποτα σχετικά δεν αναφέρει αυτή η πρόταση έκθεση. Οπότε ε, πραγματικά θα πρέπει να γίνουν μια σειρά από αλλαγέ εδώ έτσι ώστε να καταστεί πιο ισορροπημένη αυτή η έκθεση που αυτή τη στιγμή δεν είναι πραγματικά ισορροπημένη και ελπίζω πραγματικά η συγκέντρια να είναι σε θέση να είναι διατεθειμένη να γνωρίσει και εκείνα τα στοιχεία ε, τα οποία θα μπορούσαν πραγματικά να βοηθήσουν τι ε, λιγότερο αναπτυγμένε περιοχέ αντί συνέχεια να ασκεί κριτική στην δημοσιονομική πολιτική. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο, κύριο Ρόπ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Δεν μπορούμε να δρανίσουμε, πρέπει να συνομιλήσουμε για αυτές τις υστερούσες περιοχές, τις περιοχές με χαμηλό εισόδημα. Διαφορετικά, οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα ε, θα κινηθούν ανεξέλεκτα. Το κεφάλαιο πηγαίνει προς τις πιο πλούσιες χώρες και το εργατικό δυναμικό κινείται προς τις πιο πλούσιες χώρες και έτσι ε, δημιουργούνται προβλήματα για τις περιοχές. Και αν δεν βρούμε μακροχρόνιες λύσεις, δεν θα είμαστε σε θέση να πετύχουμε και πολλά πράγματα. Αυτό φοβάμαι. Οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών φτάνουν μέχρι και πέντε φορές την κατάσταση, μέση κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές λοιπόν μεταξύ περιοχών. Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα. Ε, σε ποιες λύσεις μπορούμε να καταλήξουμε για να καλύψουμε τα κενά να μειωθούν οι διαφορές. Χαίρομαι που η έκθεση αναφέρεται στον περιορισμό των μακροοικονομικών ερησιμοτήτων. Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα και θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τα ριζικά αίτια της ειστερήσεως αυτών των περιοχών. Και εγώ βλέπω, εγώ ίδιος κάποιους λόγους ανεπαρκή διοικητική, διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία των Δήμων και έλλειψη οικονομικών πόρων, κυρίως σε μικρές περιοχές, παραμεθόριες περιοχές και πιστεύω ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να εμπιστευθούν περισσότερο την τοπική τους αυτοδίκηση. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να καθορίσουν στόχους μεν, αλλά η τοπική αυτοδίκηση θα πρέπει να έχει επαρκή αυτονομία ώστε να βρίσκει τις βέλτιστες λύσεις για την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί. Αυτό μπορούμε να το πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να κολλάμε στις λεπτομέρειες. Αυτό που αποτελεί λύση στη Φιλανδία δεν είναι απαραίτητα λύση για την Κύπρο. Θα πρέπει να σκεφτούμε ποιε είναι δανειοδοτικέ, δανειοληπτικέ μάλλον δυνατότητε που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση των διαφορών χωρών. Και η μακροοικονομική αιρεσιμότητα είναι ένα εμπόδιο εδώ. Διότι όταν χρηματοδοτούνται προγράμματα, πρέπει να διατεθούν και οι κατάλληλοι πόροι. Και οι δήμοι χρεώνονται και δεν μπορούν να επενδύσουν σε έργα και προγράμματα όσον αφορά το διοικητικό δυναμικό. Όταν μια χώρα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι έχει επαρκέ διοικητικό δυναμικό, θεωρητικά. Στην πράξη όμω αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Σε κάποιε περιοχέ, σε πολύ μικρού δήμου, βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη ε, διοικητικού δυναμικού. Χρειάζεται κάποια συμβουλευτική αρρωγή, χρειάζεται συμπληρωματική χρηματοδότηση, κατάρτιση για τη διοίκηση της τοπικής αυτοδιοίκησης διότι πολλά εξορτώνται από το πώς λειτουργούν οι δήμοι και οι κοινότητες. ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια για την πρώτη αναφορά. Θα σταθώ στην έκθεση της Επιτροπής. Συμφωνώ εν μέρη με την όλη διάγνωση στην οποία προβαίνει και που εντοπίζει πέντε αίτια που δημιουργεί την αναπτυξιακή στέρηση των περιοχών. Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών με τις σχετικές μακροοικονομικές ανισορροπίες που θέτουν σε κίνδυνο ε, την πολιτική συνοχή, το πολύ χαμηλό επίπεδο της απασχόλησης, το πολύ χαμηλό επίπεδο ανθρώπων που έχουν ολοκληρήσει ανώτερη εκπαίδευση, ανώτερη εκπαίδευση, δεν έχει αναπτυχθεί έρευνα και ανάπτυξη και δεν υπάρχει μεγάλη σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και χώρου εργασίας και λόγω διοικητικών διοικητικού προβλήματος και ξεπερασμένου διοικητικού συστήματος, μαζική μετανάστευση κυρίως των νέων που ήδη έχουν εκπαιδευτεί και έχουμε μείωση του πληθυσμού ολόκληρων περιοχών και δημιουργείται κενό δημογραφικό και έλλειψη δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, πτώση τους. Και εγώ δεν συμφωνώ με τις λύσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυση της σύνδεσης με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ε, της πολιτικής συνοχής και των διαθωτικών μέτρων, κυρίως για το χώρο εργασίας. Έχουμε δεκάδες ε, συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα με τα χρόνια. Πρέπει να εξηγήσουμε άπαξ διάπαντος στους πολίτες ποιες είναι οι διαθωτικέ μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται. Διότι ε, μέχρι τις μηδενικές κυρώσεις που επευλήθησαν στην Ισπανία και την Πορτογαλία πρέπει να επιμείνουμε με το διάστημα 23 όσον αφορά τους μηχανισμούς ε, κυρώσεων. Λοιπόν, τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις μεταρρυθμίσεις διαθωτικές. Πώς τις εννοεί, όπως δηλώνουν οι Επίτροποι και ιδιαίτερα ο κ. Ντομπρόσκης, μεταρρύθμιση αγοράς εργασίας, παρεμβάσεις όσον αφορά την υγεία, τις συντάξεις, ιδιωτικοποίησεις. Εκεί δεν συμφωνούμε. Άλλο όμως είναι οι επενδύσεις για την εκπαίδευση, να αυξηθεί ε, ε, η ελκυστικότητα μιας χώρας, να μένουν οι νέοι εκεί. Ε, μετά η καταπολόμηση της φοροδιαφυγής, η ενίσχυση των στρατηγικών ε, φιούς εξειδίκευσης, η μείωση του κενού που υπάρχουν μεταξύ υποδομών σε κάποιες περιοχές όπου έχουμε ακόμα ε, απερχιωμένη προσέγγιση. Χρειάζεται επίση τεχνική αρρωγή, ώστε να ισχυθεί η δυνατότητα που έχουν τα κράτη-μέλη στη δίκηση για τη χρήση σωστή των κοινοτικών πόρων. Χρειάζεται επαρκή ε, εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα τη δίκηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ανάλυση και εφαρμογή των κανόνων των διαθετικών ταμείων σε επενδύσει. Υποστηρίζουμε οποιαδήποτε δράση που οδηγεί στο να ξεπεράσουμε τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα ε, και να έχουμε νέο, πάρα πολλού νέου κανονισμού. Χρειάζεται αναθεώρηση της ρήτρα περί επενδύσεων, ώστε οι επενδύσει σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο που συγχρηματοδοτούνται μέσω των διαφόρων ταμείων να εξαιρούνται μέσω των εθνικών ε, περιφερειακών προσεγγίσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Συμφωνούμε με ο καθορισμό των μεταρρυθμίσεων των διθωτικών που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν ε, Θα πρέπει θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι φορείς της προσπάθειες. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι είχε γίνει με την έκθεση Westphal όσον αφορά το μέλος πολιτικής συνοχής. Εμείς θα φτάσουμε μέχρι την, ε, την Ολομέλεια που υπάρχουν διαφορετικές ισορροπίες με κάποιες ε, τροπολογίες οι οποίες ε, προσπίζονται την πολιτική της συνοχής. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των πολιτικών δυνάμεων. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει άλλος που να ζητά το λόγο από τα μέλη της Επιτροπής των περι, ε, περιφερειακής ανάπτυξης. Θα δώσω το λόγο στον κ. Τέξτρα που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Yes. Thank you for the floor. I wanted to... Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα εντάχει να απαντήσω σε ζητήματα που εφήγησαν και σχόλια. Θα ήθελα να πω ότι το ε, έγγραφο εργασίας της Επιτροπής συνετάχθη για λόγους ανάλυσης και αφορούσε διάφορα τμήματα της, ε, Επιτροπή, της Ευρώπης και περιφέρειες και δεν είχε στόχο να χρησιμοποιηθεί για την κατανομή ε, χρηματοδότησης. Ως προς την πολιτική συνοχής μετά το 2020 δεν θέλουμε να υπάρχουν προσκόμματα ως προς ε, ε, πολυπεριφερειακές ε, χρηματοδοτήσεις. Θεωρούμε ότι και άλλοι δείκτες είναι σημαντικοί για ανάπτυξη στρατηγικής και για τον ορισμό προτεραιοτήτων στις διάφορες περιφέρειες και θεωρώ ότι ο δείκτης περιφερειακής προόδου είναι πολύ σημαντικός, θα επικαιροποιηθεί το 2019. Ε, συνετάξαμε αυτή την έκθεση για να δούμε πώς εξελίσσονται αυτές οι περιφέρειες και θα συνεχίσουμε το, την εποπτεία αυτών των περιφερειών έτσι ώστε να μπορέσει να τις ε, συνδράμει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω πολιτικής ε, συνοχής. Η έβδομη εκθεση συνοχης οριζει οτι η το Ταμείο Συνοχής είναι ένα βασικό επενδυτικό μέσο και τονίζουμε και το ρόλο της διακυβέρνησης. Υπάρχει ένα κεφάλαιο στην έκθεση συνοχής και προβάλλουμε σχέδια επενδύσεων για να αναγνωρίσουμε που στο σημείο στην πολιτική διακυβέρνηση ε, χρειάζονται βελτιώσεις. Δηλαδή η έκθεση επιχειρήσεων μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα για παράδειγμα για να δούμε πού υπάρχουν προβλήματα στις κυβερνητικέ πολιτικές. Καθώς και η έκθεση για το επιχειρήν ως προς την μακροοικονομική πολιτική. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πρόωρο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δηλώσει το οτιδήποτε. Κυρία Τζουφρίντα, θα θέλατε να απαντήσετε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήμουν σίγουρη ότι η έκθεση θα οδηγούσε στα ενδυμικά αποκλίνοντα στοιχεία της Επιτροπής μας. Ε, το ήξερα ότι δεν ε, υπάρχει κοινή προσέγγιση και αυτό φαίνεται και από ορισμένα σημεία που ανέφεραν οι συνάδελφοι. Νομίζω όμως ότι όταν αναθεωρηθεί η πολιτική συνοχής θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μία αίσια έκβαση. Είμαι πεπισμένη ότι η έκθεση θα πρέπει να την χάνει πολιτικής προσέγγισης, διότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να λάβει θέση για τις ε, προτάσεις ως προς προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαίρομαι διότι εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε το 2019 θα έχουμε νέους ε, δείκτες, ε, τους οποίους θα λαμβάνει υπόψη η Επιτροπή που χρειαζόμαστε φυσικά για να προσαρμόσουμε τις πολιτικές συνοχής και όλα τα συμπαρομαρτούντα κάτι το οποίο χρειάζεται αυτή την επικαιροποίηση σε σχέση με τη συνετή προσέγγιση που προαναφέρθηκε. Συμφωνώ με τον συνάδελφο, αλλά θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι αυτή η συνετή προσέγγιση στο εγγύς παρελθόν δεν οδήγησε σε αποτελεσματικές λύσεις ιδιαίτερα όταν ε, υπήρχε μια έκτακτη κατάσταση ιδιαίτερα, όταν μιλάμε για περιφέρειες με αναπτυξιακή καθυστέρηση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα καθαρά κυρωτικό πλαίσιο, διότι όταν δρά κανείς επιγόντως, σε περιπτώσεις κατεπίγουσας ανάγκης, δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι αντιδρούμε σωστά. Θα πρέπει να θέσουμε λύσεις επί χάρτου τη στιγμή που υπάρχουν περιφέρειες ε, που χρήζουν της ε, πολιτικής συνοχής. Και αυτό είναι και ο απότερος στόχος της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει να βρούμε ένα σημείο εξισορρόπησης, όλοι συμφωνούμε επ' αυτού, και θα ήθελα να υπενθυμίσω σε άλλους συναδέλφους ότι οι πολιτικές λιτότητας αυτές τις περιφέρειες ενθαρρύνουν τις περικοπές δημοσίων επενδύσεων. Κάτι το οποίο ε, οδηγεί μόνο στην ε, αποπληρωμή του χρέους και σε τίποτα άλλο. Και θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μία αναπτυξιακή πορεία προς ε, δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή εξισορρόπηση, κάτι το οποίο όμως ε, σημαίνει ότι δεν θα πρέπει, θα πρέπει να μπλοκάρουν τις χρηματοδοτήσεις τα κράτη-μέλη ως προς τη διακυβέρνηση θα πρέπει να βελτιωθεί στα κράτη-μέλη, στο εσωτερικό των κρατών μελών και συγκεκριμένων περιφερειών, αλλά αυτό είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε την πολιτική συνοχής, ιδιαίτερα στις περιφέρειες με αναπτυξιακή καθυστέρηση. Αυτό είπε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, δηλαδή ο, γίνονται ασκήσεις κατανομής, αλλά δεν θα πρέπει να δεσμεύουν τις περιφέρειες σε μια πολύ αυστηρή ε, ταξινόμηση. Γι' αυτό Ελπίζω ότι θα βρούμε ένα σημείο συνάντησης και εξισορρόπησης με τις τροπολογίες συμβιβασμού. Γιατί όπως είδαμε και στις προγενέστερες εκθέσεις, αυτός είναι ο απότερος στόχος. Πρέπει να προβούμε σε επιλογές μέσα στα πλαίσια της έκθεσης και συμπεραίνω, ολοκληρώνω γιατί βλέπω ότι ήρθε η Επίτροπος, η κυρία Κρέτσου και θα πρέπει να φτάσουμε σε μία αγαστή συνεργασία με την Επιτροπή. Μιλάμε για κοινούς στόχους έτσι ώστε η πολιτική σύνοχης να είναι αποτελεσματική για να βοηθήσουμε τις ε, περιφέρειες σε ύφαση. Αναμένω τις τροπολογίες σας και πιστεύω ότι θα έχουμε μια επικοδομητική ε, συνάντηση και καλωσορίζω και την Επίτροπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ενημερώσω λοιπόν πως η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών σε σχέση με αυτή την έκθεση είναι η 14η Δεκεμβρίου το μεσημέρι. Στις 12 το μεσημέρι. Και στη συνέχεια η ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή μας θα λάβει χώρα το Φεβρουάριο. Επαναλαμβάνω, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 14 Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή τη συζήτηση. Κλείνουμε με την ε, με αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρης σας διαταξής μας ε, και βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση για να καλωσορίσω την Επίτροπο Κρέτσου για μία ακόμα φορά στην Επιτροπή μας. Εδώ λοιπόν στο κείμενο που έχω μπροστά μου αναφέρεται ότι η Επίτροπος μας έχει επισκεφθεί έξι ε, φορές ε, προηγουμένω φέτος στην Επιτροπή μας, οπότε επιχαίρουμε το γεγονό ότι έχουμε τη δυνατότητα να συζητούμε τόσο συχνά με την Επίτροπο όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά για την Επιτροπή μας. Ε, την... Καλωσορίζω λοιπόν εδώ σήμερα και α, δίνω α, το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε και πάντοτε ε, χαίρομαι όταν βρίσκομαι εδώ. Αξιότυπα λοιπόν μέλη αυτής της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, όπως είπα, με χαρά μου βρίσκομαι εδώ και θα ήθελα ε, εν συντομία να σας ενημερώσω σε σχέση με το πακέτο το οποίο εγκρίθηκε χθες σε ό,τι αφορά ε, την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε στην ίδια την πολιτική συνοχής. Όπως Ίσως ε, όλοι θα παρακολουθήσατε λιγότερο ή περισσότερο τις ε, παρουσιάσεις εχθές. Θα ε, γνωρίζετε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πακέτο και μάλιστα σε σχέση με τρεις πτυχές. Ε, δηλαδή το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το περιεχόμενο του πακέτου είναι ε, πολύ ευρύ και ε, καλύπτει μια σειρά από σημαντικές ιδέες. Αλλά επιτρέψτε μου εγώ να περιοριστώ στις πιο σημαντικές από αυτές. Καταρχήν η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου έτσι ώστε να παρέχει υποστήριξη σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέρχονται δύσκολες περιόδους όπως είχε κάνει δηλαδή και ο πολιτικός, μηχανισμός σταθερότητας η δικλίδα, αν θέλετε, αυτή ασφαλείας του Ταμείου θα επιτυγχάνεται μέσω των συνθηκών της Ένωσης, όχι δηλαδή μέσω διακυβερνητικής συνεργασίας. Με αυτόν τον τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να παίξει ένα ισχυρότερο ρόλο στη λειτουργία, ε, για τη λειτουργία και την παρακολούθηση αυτού του Ταμείου. Δεύτερο, η ολοκλήρωση της ε, συμφωνίας σε ό,τι αφορά την ε, σταθερότητα, ε, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση, στο πλαίσιο ακριβώ πάντοτε τη Ένωση. Και πάλι εδώ έχουμε καλέ ειδήσει για το Κοινοβούλιο και για τη Δημοκρατία, γιατί ακριβώ θα σημάνει περισσότερη ανάληψη ευθυνών και περισσότερη αποτελεσματικότητα. Ε, και μετά σε ό,τι έχουμε τα νέα ε, εργαλεία, του χρηματοδοτικά εργαλεία του προπολογισμού, δηλαδή σε ό,τι αφορά ειδικότερα την πολιτική συνοχή με εθελοντική βάση μια ε, στρατηγική, μια διευκόλυνση ε, σύγκλησης ε, και επίσης μια εγγύηση σε ό,τι αφορά την, τον τραπεζικό τομέα αλλά και ένα τομέα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση μεγάλων ασυμμετρικών σοκ αλλά και ο διορισμός του Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομικών ο οποίος ή η οποία γιατί δεν ξέρουμε ακόμα το φίλο όταν ε, αναφερόμαστε σε αυτόν, σε αυτήν την Υπουργό Οικονομικών, θα αναλάβει χρέη την Προέδρου της Επιτροπής και ε, Προέδρου του Ευρωκρούπου. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στο πλαίσιο του μηχανισμού λήψη αποφάσεων εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, περνάω στη δική μα ε, πολιτική, πολιτική συνοχή. Όπω γνωρίζετε, κατά του τελευταίου μήνε κάναμε μακρέ συζητήσει με τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο ειδικότερα τη ε, συνεδρία του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Τα κράτη-μέλη εξέφρασαν την υποστήριξή του απέναντι στην πολιτική συνεχή και συμφώνησαν ότι θα πρέπει να παραμείνει ανάμεσα στι κύριε πολιτικέ τη Ένωση και μετά το 2020. Ε, και πράγματι χάρηκα για το γεγονό ότι όλοι ε, οι υπουργοί μα υποστήριξαν σε αυτή την ε, προσέγγιση μα και ελπίζω πω ε, και οι υπουργοί οικονομικών θα μα υποστηρίξουν με τον ίδιο τρόπο. Τα δικά μου επιχειρήματα βέβαια βασίστηκαν ήδη στα επιτεύγματα τη πολιτική συνοχή μέχρι τώρα, τα οποία κατά τελευταία μου επίσκεψη εδώ στην Επιτροπή σα τα παρουσίασε. Δηλαδή, η κρίση άφησε μεγάλε σουλέ στον οικονομικό, κοινωνικονομικό ιστό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη από ένα στα κράτη-μέλη, ώστε να είναι πιο ανθεκτικά απέναντι στην ε, παγκοσμιοποίηση και ε, στη βιομηχανική μεταβολή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε καλύτερα του τομεί εκείνου στου οποίου μπορεί να έχει πραγματικό αντίκτυπο η πολιτική συνοχή. σω δηλαδή τα υφιστάμενα πλαίσια να είναι υπερβολικά άκαμπτα, να θα πρέπει να γίνουν ε, πιο προσαρμόσιμα, έτσι ώστε να εστιάζουμε σε νέου τομεί προτεραιότητα και περισσότερο στα αποτελέσματα. Όπω αναφέρθηκε και στην έκθεση, το χαμηλό επίπεδο διακυβέρνηση και οι διαστροτικέ αδυναμίε μπορούν να αποτελέσουν αποτελέσουν εμπόδιο σε ό,τι αφορά τι δημόσιε επενδύσει. Η πολιτική συνοχή δηλαδή δεν μπορεί να είναι αυτή Θα πρέπει να υποστηρίζει και να υποστηρίζεται από σημαντικέ διαφορετικέ μεταρρυθμίσει. Ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να παρέχουμε τα κατάλληλα κίνητρα για ε, αυτέ τι μεταρρυθμίσει. Ε, πέρα τη συνεδρία του Συμβουλίου των Γενικών Υποθέσεων, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα δύο σημαντικά έγγραφα. Καταρχήν την ανακαίνωση σε ό,τι αφορά τι συνοριακέ περιοχέ τη Ένωση που καλύπτει και ζητήματα πέραν τη χρηματοδότηση. Ένα από τα νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται εκεί είναι τα border focal points, ε, τα οποία θα, ε, ή ένα border focal point, το οποίο αποτελεί τα περιεχόμενα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει υποστήριξη στα κράτη-μέλη ε, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση εμποδίων νομικού αλλά και διαχειριστικού χαρακτήρα στα σύνορα. Με αυτόν τον τρόπο, στο πλαίσιο δηλαδή αυτή τη ομάδα, θα υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγή απόψεων. Επίση, τον Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά τη διαπεριφερειακή συνεργασία, ε, προβήκαμε σε ε, ε, ένα πολιτικό έργο και την προκήρυξη εξήλωση αναφέροντο σε ό,τι αφορά εταιρικέ σχέσει από του κλάδου τη μηχανία, ακαδημαϊκού κλάδου και ούτω καθεξή. Και παρά την πολύ σύντομη προθεσμία που είχαμε θέσει, υπήρξε καλή ανταπόκριση σε αυτή την προκήρυξη εκδήλωση ενδιαφέροντο και την επόμενη εβδομάδα θα δημοσιευθούν και όσοι κέρδισαν σε αυτό το διαγωνισμό. Η ανάδοχη δηλαδή του πιλωτικού προγραμματό. Επίση. Ε, υπήρξε δημοσίευση της ε, πριν από μερικές εβδομάδες και ε, μετά από ένα ε, μόνο χρόνο από τη χάραξη ήδη έχει ξεκινήσει αυτό το αστικό θεματολόγιο, έχουν δηλαδή ξεκινήσει εταιρικέ σχέσεις και το, ο προπολογισμό θα έχει οριστικοποιηθεί μέσα ε, στο τέλος αυτού του, έως τα τέλη αυτού του έτους. Ε, προφανώς με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ήταν αποφασιστική τα καταφέραμε όλα αυτά και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό. Επίσης η έκθεση για την αστική πολιτική έχει καταδείξει ότι η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση έπαιξε σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για τις αστικές περιοχές και πέρσι εγώ στο Γιώτο είχα τη δυνατότητα να αναφερθώ στην εφαρμογή της αστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως ανέφερα και την προηγούμενη εβδομάδα στο Ρότερνταμ, θα πρέπει να είμαστε περήφανοι και για το Cities Forum. Ε, ε, δηλαδή, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκεί εγκαινιάσαμε μια νέα συμβουλευτική ε, υπηρεσία η οποία μπορεί να βοηθήσει τις πόλεις να προβούν στις μεταρρυθμίσεις του ταχύτερα. Θα έχει την ονομασία Ούρμπης και θα δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους και τις κοινότητες να λαμβάνουν ταχαίως καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις. Επίσης, ό,τι αφορά τη στρατηγική έκθεση για την αξιοποίηση ε, των διαθροτικών ταμείων, να σα πω ότι θα δημοσιευθεί την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά μπορώ από τώρα να σας πω ότι είναι πολύ καλά τα νέα, δηλαδή η εφαρμογή έχει κινηθεί καλά ε, μέσα στο τελευταίο έτος ε, και αυξάνεται όλο και περισσότερο. Ε, έχουν επιλεγεί ε, έργα της ε, τάξης των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή ανέρχονται στο 45% της συνολού της χρηματοδότησης. Η επιλογή αυτών των project, αυτών των έργων, με την περίοδο 2007-2013 παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε καθυστερημένα η εν λόγω περίοδος χρηματοδότησης. Ε, και η εφαρμογή νέων μέτρων όπως η εκ των προτέρων ερσιμότητας ε, έχουν εφαρμοστεί κανονικά, έχουν τρέξει κανονικά. Και μετά από τη δημοσίευση, την ερχόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο θα έχω τη δυνατότητα να σε ενημερώσω περαιτέρω σε σχέση με το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης. Αλλά όσοι δεν θα παρευρεθείτε εκεί, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά και σίγουρα το 2018 μας περιμένει πολλή δουλειά, οπότε ελπίζω όλοι να έχουμε την απαραίτητη ενέργεια και να κτίσουμε λίγο τις δυνάμεις μας ε, στο πλαίσιο των διακοπών, των χριστουγεννιάτικων διακοπών και αναμένω τώρα τα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Επίτροπε. Θα ακούσουμε τις ερωτήσεις. Θα ακούσουμε τους συντονιστές, αρχίζοντας τον κύριο Βανίστελ Ρόι. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντική αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές γύρω μας. Θα πρέπει να μας πληροφορήσετε για τις αλλαγές. Θα αναφέρω ένα-δύο σημεία και θα ζητήσω για τον Αριμό να πει ένα, είναι ο μόνιμος εισηγητής για την Ελλάδα να πει κάτι και μετά για το ΣΕΦ, το Μέσο και Διασύνδεση της Ευρώπης. Ο συνάδελφος Νοβακόφ θα μιλήσει αργότερα γι' αυτό. Πρώτο σημείο. Βλέποντας και αποτιμώντας τι έγινε μετά τους κυκλώνες στο Σεν Μάρτιν Έγινε καλή συζήτηση στην Ολομέλεια. Δεν καταλήξαμε σε ψήφισμα όμως. Μας ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι και τα δύο τμήματα του, της νήσου θα αντιμετωπιζόταν ισότιμα. Από τις πληροφορίες που συλλέγουμε βλέπουμε ότι συμβαίνουν λιγότερα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Ανασυγκρότησης, συγκρίνοντας το γαλλικό τμήμα, βλέποντας τι γίνεται στο γαλλικό τμήμα, το Ταμείο Αλληλεγγύης. Δεν βλέπω πρόταση για τον, ε, την ίσο της, ε, του Αγίου Μαρτίνου. Θέλω να συνεργαστούν οι δύο χώρες. Ο κύριος Γιούνκερ τον έφερε σε επιστολή του ότι χρειάζεται κοινή προσέγγιση. Η Επίτροπος θα ήθελα να με ενημερώσει για την κατάσταση στο Σεν Μάρτενς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γαλλικά χρήματα που δεν απορροφήθηκαν για το πρόγραμμα ανοικοδόμησης του νησιού. και έχουμε στο ακροατήριο εκπροσώπους του νησιού. Δεύτερο ερώτημα. Σήμερα συζητήσαμε πώς οι διαφθορτικές ε, μεταρρυθμίσεις εφαρμόζονται. Έχει αλλάξει ο κανονισμός και ο δικός μας κανονισμός. Και τι βλέπω. Ότι το Κολέγιο των Επιτρόπων είπε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ε, τις επιδόσεις για διεθνωτικές μεταρρυθμίσεις κλπ. πλήρως. Το 6% και τα 21 δις που δόθηκαν για τα κράτη-μέλη για τη βελτίωση των επιδόσεων συνδέεται με επιδόσεις των χωρών. Και ανησυχώ και θα υποβάλω σχετική προφορική ερώτηση και σχέδιο ψηφίσματος στο Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο. Ποτέ δεν μας ενημέρωσαν ότι άρχισε κίνηση προς την κατεύθυνση των επιδόσεων και τώρα αλλάζει εντελώς η κατεύθυνση. Στην έκθεσή μας ζητήσαμε ταχεία προσέγγιση. Κυρίως προς τις χώρες που έχουν επιδόσεις. Και τώρα είναι σαν να μας κλέψανε τα χρήματα το βράδυ. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, ένα σχόλιο θετικό από το γραφείο σας και στη συζήτηση εδώ, ανταλλαγή απόψε με τα κράτη-μέλη, με τα εθνικά κοινοβούλια, άκουσα να λέτε ότι θα ελέγξετε γραμμή προς γραμμή τον κανονισμό. Να δείτε τι μπορεί να αφαιρεθεί, τι θα μείνει και τι μπορεί να αλλάξει. Θέλουμε αυτό να το συνδυάσουμε με την έβδομη έκθεση συνοχής. Να έχουμε έτοιμα τα δικά μας αποτελέσματα. Και το δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ατύπως να κινηθεί και τον Απρίλιο στην Ολομέλεια να σχολιάσει τις απόψεις μας. Να, να εξετάσει τις απόψεις μας. και να υποβληθεί κάποια πρόταση ε, πριν τις εκλογές του 2019. Ευχαριστώ κύριε Βανίστολου. Ε. Έχω τη χαρά να καλωσορίζω τους φιλοξενούμενους μας από το Σεν Μάρτεν. Είναι φιλοξενούμενοι σας, αλλά είναι φιλοξενούμενοι της Επιτροπής μας. Τους καλωσορίζω λοιπόν. Καλώς ήρθατε στην συνεδρίασή μας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και την απάντηση της Επιτρόπου όσον αφορά την κατάσταση στην είσοδο του Αγίου Μαρτίνου η κυρία Κρέα έχει το λόγο. Σας ευχαριστούμε θερμά κυρία Επίτροπε για το γεγονός ότι πραγματικά πάντοτε είστε διατεθειμένοι να παρευρεθείτε εδώ ε, και να συνεργαστείτε με τη δική μας ε, Επιτροπή. Ε, θέλω λοιπόν να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία της παρουσίας σας σήμερα εδώ έτσι ώστε να θίξω ορισμένες πτυχές αυτής της πρότασης για το EMU, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. αυτό που είπε ο κύριος Λάμπερτ νομίζω πως είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, άκουσα και εγώ με μεγάλη μου έκπληξη ε, ότι αυτό το performance reserve ε, το οποίο δεν ήθελε ε, σε καμία περίπτωση η Επιτροπή είναι κάτι το οποίο τώρα θεωρείται ως εκτιτήριο επιτυχίας. Ε, δηλαδή αποτελεί και τμήμα του εθνικού φακέλου για, τους, ε, για τα κράτη-μέλη, οπότε με εκπλήσει τώρα ε, το γεγονός ότι πρόκειται να επενδυθεί, να αφοσιωθεί αυτό το αποθεματικό στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα ή όχι. Αλλά νομίζω πως αποτελεί μία πλήρη αλλαγή πορείας. Δηλαδή πριν από τρία ή το πολύ τέσσερα χρόνια η Επιτροπή ήθελε ακριβώς το πολυ τεσσερα χρονια Οπότε διαρωτώ με λίγο. Μετά, σε ό,τι αφορά το SSP. Ε, και εδώ ο κανονισμό ε, υποτίθεται πω θα αλλάξει για να υπάρχουν περισσότερα κονδύλια και ούτω καθεξή. Ακούω με χαρά μου ότι πράγματι λειτουργεί καλά το εν λόγω εργαλείο και ίσω καλό θα ήταν να λάβουμε κάποια σχετικά στοιχεία. Αλλά Επιτρέψτε μου και σε σχέση με αυτό να εκφράσω την έκπληξή μου, γιατί στο πλαίσιο του τριμερού διαλόγου που έγινε πρόσφατα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία Omnibus, εμεί καταφέραμε να επιβάλλουμε ένα πακέτο διαφάνεια ορατότητα, ένα visibility package, και μέσω του οποίου ζητήσαμε από την Επιτροπή ε, κάποια κονδύλια τη τεχνική βοήθεια, του technical assistance, σε ορισμένο ποσοστό να αξιοποιηθούν για την καλύτερη ορατότητα, την καλύτερη προβολή αυτή τη πολιτική πράγμα που και εγώ θεωρώ απαραίτητο, αφού ακόμα και σήμερα πολλέ πολίτε και πολλοί πολίτε δεν γνωρίζουν τι ακριβώ συμβαίνει ε, στα κράτη-μέλη του, ε, ε, πώ δηλαδή τα βοηθάει και στι περιφερειέ του η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν αναφέρθηκε ότι δεν μπορεί να υπερβεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό αυτή η χρηματοδότηση, γιατί ακριβώ. Ε, δεν ε, μπορεί να στερηθεί περαιτέρω κονδύλια από την τεχνική αρρωγή η Επιτροπή. Αλλά μόλι τώρα ακούσαμε ότι 300 εκατομμύρια ευρώ συμπληρωματικά θα βγουν από την τεχνική βοήθεια. Άρα τελικά θα είχαν υπάρξει περαιτέρω κονδύλια που θα μπορούσαν να είχαν βγει προηγουμένω από την τεχνική βοήθεια για να πάνε εκεί. Οπότε ε, δεν έγινε κάποιο καλό συντονισμό. Αν μπορούμε να καταφέρουμε και τα δύο, έχει καλό, Αλλά πραγματικά θα πρέπει λίγο να το ξανασκεφτούμε. Δηλαδή θα πρέπει ε, να γίνονται τα βήματα το ένα μετά το άλλο. Στο πλαίσιο δηλαδή του κανονισμού Omnibus είχαμε θέσει εμεί πολύ συγκεκριμένε προτάσει. Μήπω λοιπόν θα είναι δυνατόν να γίνει ένα συνδυασμό ε, αυτών των δύο ε, μέτρων. Εν πάση περιπτώσει, ίσω εγώ κάτι μπορεί να μην κατάλαβα σωστά σε ό,τι αφορά δηλαδή, το πώ ακριβώ θα λειτουργήσει το νέο εργαλείο SSP. σω να μην λάβαμε και όλε τι προφορίες δηλαδή από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Σω θα μπορούσατε να κάνετε και κάποια σχόλια από την πλευρά σας Επιτροπή σε σχέση με αυτό. Ευχαριστώ. Thank you very much, Thomas. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μασίτς, κυρία Τάμασίτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη, πώς μπορούμε να επηρεάσουμε μελλοντική νομοθεσία που θα προωθεί περισσότερα πολυταμιακή χρηματοδότηση και ποιες προϋποθέσεις θα πληρούν τα κράτη-μέλη για καλύτερη εφαρμογή της πολυταμιακής χρηματοδότησης. Και τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν αρκετά χρηματοπιστικά ε, μέσα ή διστάζουν λόγω των κινδύνων. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και να μειώσουμε τον κίνδυνο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε χώρες να δημιουργήσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για μελλοντική καλύτερη εφαρμογή των διαφόρων σχετικών προγραμμάτων. Ευχαριστώ κύριος Βαν Μίλτεμπερκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, κύριε Επίτροπε. Πάντα χαρά για μα να μπορούμε να συζητούμε μαζί σα ενδιαφέροντα ζητήματα. Είμαι κάπω πιο θετικό όσον αφορά τη χθεσινή πρόταση. Διότι αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε θετικέ μεταρρυθμίσει στην Ευρώπη, θα πρέπει να έχουμε και θετική στάση. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την προώθηση των διαθωτικών μεταρρυθμίσεων και των σχετικών προγραμμάτων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διάφορες ε, συμφωνίε, τον ισχύοντα κανονισμό, αλλά εγώ είμαι πιο ανοιχτό από ότι άλλοι συνάδελφοι ενδεχομένω να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Διότι θετικέ μεταρρυθμίσει χρειάζονται στην Ευρώπη. Με κάποιο τρόπο λοιπόν θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε τι αλλαγέ αυτέ. Δεύτερον, όπω αγαπητό συνόδελφο ο κύριο ε, Βανίστερ Ρόι αναφέρθηκε στο Σεν Μάρτιν. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ στου εκπροσώπου του Σεν Μάρτιν, τον κύριο Μπλοντέιν και τον κύριο Άρνολτ που είναι εδώ στην αίθουσα. Η καταστροφή μετά ε, το κυκλώνα ε, Ήρμα ε, σημαίνει ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Να μείνω στα λόγια, το Σεπτέμβριο ήδη έστειλα γράμμα στον κύριο Γιούνκερ και έχω την απάντηση. Και στην απάντηση αναφέρει ότι θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα κινητοποίησεω και παραθέτω συμπληρωματική, πόρη και αναφέρει επίσης ότι η Ευρώπη χρειάζεται συντονισμένη απάντηση όσον αφορά τις ανάγκες το, του λαού τη νήσου, του Σεν Μαχτέ και του Σεν Μάρτεν. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη τις νομικές διαφορές και το καθεστώς του γαλλικού και του ολλανδικού τμήματο του νησιού. Εδώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα, θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό. Δεν θα ήταν συνετό όπως έκανε η Γαλλία και έκανα η Ολλανδία να έχουν ένα εθνικό συντονιστή που θα συντονίζει ε, τις προσπάθειες ε, ε, ε στο νησί για την ανοικοδόμηση και να υπάρχει ίσως και Ευρωπαίος συντονιστής που θα συντονίζει όλες τις προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα διάφορα τμήματα και να δούμε τι είναι δυνατόν να κινητοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό από τις ισχύουσες χρηματοδοτικέ ε, δυνατότητες που προσφέρονται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα μια απάντηση. Είστε πρόθυμοι να το εξετάσετε, διότι νομίζω ότι αυτό χρειαζόμαστε Ευρωπαίο συντονιστή που πραγματικά θα προσπαθήσει να κάνει τη δουλειά του το καλύτερο που μπορεί εκείνο ή εκείνη σε στενή συνεργασία με τον Ολλανδό και Γάλλο συντονιστή στο νησί, ούτω ώστε τελικά να μείνουμε στα λόγια και να έχουμε δράση. Γιατί αυτό που λείπει είναι η δράση, αυτό χρειάζεται. Πρέπει επίση να προστατεύσουμε όλους τους πολίτες της Καραϊβικής. Μετά αναφερθήκατε στην εφαρμογή, στην υλοποίηση και ποια είναι η κατάσταση. Κάπως πιο θετικά τα πράγματα από ότι πριν από ένα χρόνο, αλλά πήγαμε στη Ρουμανία, στη χώρα σας, την επισκεφτήκαμε, τη χώρα σας, το κράτος μέλο τη και άκουσα σοβαρές διαμαρτυρίες για τη γραφειοκρατία, για την έλλειψη απορροφήσεως πόρων, ε, επίσης λόγω γραφειοκρατίας και εκεί. Από ό,τι κατάλαβα, μου είπαν οι υπηρεσίες σας ότι λόγω του 1 συν 3 του χρόνου θα αντιμετωπίσει προβλήματα σοβαρά η Ρουμανία, θα χάσει πιθανότατα τα χρήματα που τους έχουν ε, ε δοθεί, έχουν προσημειωθεί για αυτήν. Τι δράσεις προβλέπετε να ακολουθήσετε. Και εδώ θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν θα ήθελα να παραπέμψετε στην έλλειψη πρωτοβουλίων των περιφερειών που αναφέρθηκε πριν. Περιμένει η Ρουμανία κάτι τέτοιο, περιμένει ο λαός να δει πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα θετικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενώσης προς όφελός τους. Οπότε ζητώ συγκεκριμένες δράσεις. Ευχαριστώ. Καλώς. Κύριος Ράπε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την δυνατότητα να σας ξαναδούμε εδώ, να σας ξανασυναντήσουμε. Έχω κάποια, κάποιες ιδέες που ήθελα να εκφράσω, ευπρόσδεκτα αυτά που είπατε, δηλαδή ότι το νέο, το νέο πακέτο για τη συνοχή ε, θα ενισχυθεί και θα είναι πιο ευέλικτο. Θα είναι ευέλικτο μόνο για κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο ή θα είναι ευέλικτο και μέχρι το επίπεδο δήμων και κοινοτήτων. Έτσι δημιουργούνται νέες δυνατότητες, αν ισχύει αυτό. Και κάτι άλλο. Αναφερθήκατε στη χρηματοδότηση ε, προγραμμάτων στην τρέχουσα περίοδο. Είπατε ότι Ήδη έχουν επιλεγεί τα μισά προγράμματα, αλλά βλέπουμε ότι φτάνουμε στο τέλος του τέταρτου έτους. Μας μπαίνουν μόνο τρία χρόνια. Είμαστε στα μισά, ας πούμε. Και βλέπουμε ότι πιο αδύναμες χώρες, πιο αδύναμες περιοχές, λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, ότι εκεί παίρνουν 80% των επενδύσεων από χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε 3-4 χρόνια θα αυξηθεί η ροή των χρημάτων, αλλά θα αυξηθεί και το κόστος. Δεν πιστεύετε ότι στο μέλλον θα έπρεπε να προβλέψουμε διαφορετικό μηχανισμό, ούτω ώστε η απορρόφηση των πόρων να γίνεται πιο ομαλά, χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις. διασυνοριακή συνεργασία με τρίτες χώρες. Προβλέπετε κάποια νέα πρότυπα να εφαρμοστούν στο μέλλον. Η συνεργασία θα είναι παρόμοια, θα αλλάξει. Άλλη μια ερώτηση. Αφορά την κοινή αγροτική πολιτική. Δεν θα πρέπει να συμβάλλει αυτή και αυτή η πολιτική στη συνοχή και να μειώνει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ ε, διαφόρων περιφερειών. Κύριε Νταμάτο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επίτροπο που είναι εδώ μαζί μας για άλλη μία φορά για να συνοψίσω ορισμένα καυτά ζητήματα όπως ε, όρισε το κίνημα των πέντε αστέρων κατά της ε, μακροοικονομικής ερεσιμότητας, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει λανθασμένη επέμβαση του συντάξεις, στα εργασιακά και ούτω καθεξής. Έχουμε πληγή από φυσικές καταστροφές, αλλά δυστυχώς ε, δεν υπάρχει πλήρης ανταπόκριση, άμεση ανταπόκριση. Πρόκειται για φυσικές καταστροφές που συνεχώς επισυμβαίνουν όλο και περισσότερο στην Ευρώπη αν και γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο πρόσκομα είναι το Συμβούλιο, θα ήθελα να μην παρετηθείτε. Πότε μπορούμε να αναμένουμε μία στοχοθετημένη πρόταση με μεγαλύτερη ευελιξία, περισσότερη, μεγαλύτερη κατανομή πόρων και ε, συγκεκριμένες προκαταβολές γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει το όριο των 30 εκατομμυρίων. Υπάρχει και η οδηγία Omnibus. Φαντάζομαι ότι θα γίνουν και νέες ρυθμιστικές προτάσεις το Μάιο-Ιούνιο του 2018. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία αλλά και συμμετοχή των πολιτών ήδη από τώρα, πριν από τα λειτουργικά προγράμματα. Ξέρετε ότι ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Εταιρικότητας εφαρμόστηκε τύπης χωρίς τη συμμετοχή των οικονομικοκοινωνικών φορέων και χωρίς έγκαιρη προσέγγιση και προσβασιμότητα, ιδιαίτερα για τις ΜΚΟ και τους κοινωνικούς φορείς η εξάντε αιρεσιμότητα, δηλαδή ένας δεσμευτικός μηχανισμός που ορίζει τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων σε αυτή την εταιρική σχέση, καθώς και τα ε, εταιρικά περιφερειακά προγράμματα αποτελούν μία απτή πραγματικότητα. Θα πρέπει να υπάρχει μία πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που να αφορά όλους τους πολίτες. Τι περιμένετε εσείς από αυτό. Μπορούμε να έχουμε τη δημόσια δέσμευσή σας ότι θα δεσμευτείτε γιατί οι πολίτες συμμετέχουν και θέλουν να συμμετέχουν έτσι ώστε να υπάρχει μια συνεργατική πολιτική που να βρίσκεται πολύ κοντά στις περιφέρειες. Έχω τρία ονόματα ακόμα. Ο κύριος Νοβάκοφ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Επίτροπο Κρέτσου γιατί κατέβαλε μεγάλες ε, προσπάθειες να επισκεφτεί όλες τις χώρες που υπέστησαν φυσικές καταστροφές ε, μεταξύ αυτών και την ε, Πορτογαλία, γιατί έχει σημασία να προβάλλουμε ένα ανθρώπινο πρόσωπο της κρίσιμες στιγμές. Θα ήθελα να εκφράσω ορισμένες ανησυχίες. Καταρχήν με την χτεσινή ανακοίνωση της Επιτροπής, γιατί θα αλλάξει τον τρόπο χρηματοδότησης του SPR. Είμαι πεπισμένος ότι υπάρχουν καλές προθέσεις, αλλά θεωρώ ότι οι πολιτικές συνοχής ε, ε, περιβάλλονται από άλλα. Στην αρχή είχαμε ε, την ταχεία προσέγγιση με τα fast tracks, μετά το ΣΕΠ, το Ταμείο Συνοχής και τώρα μιλήσαμε για συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. θεωρούμε ότι θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τις διάφορες πτυχές της ε, πολιτικής συνοχής. Ίσως φαίνεται ότι περιστοιχίζεται καλά η πολιτική, αλλά δεν θα πρέπει να παρετηθούμε από τα κεκτημένα. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι το τι μας περιβάλλει και πάντα μπορούμε να βρούμε συμμάχους. Γιατί αν αλλάξουμε τώρα τους κανόνες του παιχνιδιού, ιδιαίτερα ως προς τις αποδόσεις, ε, τότε θέλουμε να ε, αποδώσουν τα κράτη-μέλη, αλλά αλλάζουμε τους κανόνες εν μέσω παιχνιδιού γιατί θέλετε να αποδομήσετε ένα σπίτι και να χρησιμοποιήσετε τα τούβλα για να χτίσετε ένα διαφορετικό. Επίσης, βρισκόμαστε έξι μήνες πριν από την εφαρμογή του νέου κανονισμού. Και έχουμε τουλάχιστον δύο προτάσεις κανονισμού σε σχέση με την πολιτική συνοχής. Φοβάμαι το τι θα συμβεί το επόμενο εξάμεινο χαίρομαι διότι θα μας ε, δώσετε περισσότερες αποσαφηνήσεις γιατί προσπαθώ να βρω θετικότερα σημεία για τη χρήση των 21 εκατομμυρίων γιατί γίνεται λόγος για μέρος ή το όλων για τις διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις. Εάν είναι τόσο κρίσιμο για το Σύμβουλιο, τότε θα πρέπει να βρούμε φρέσκο χρήμα για τη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαρέμον έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρόμαστε γιατί βρισκόσαστε ενώπιόν μας με τέτοια συχνότητα. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Είπατε ότι θα δημοσιευτεί μία έκθεση για την εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων και τα έκτακτα μέτρα υπέρ της Ελλάδας. μέσα στα πλαίσια των ε, δύο τελευταίων δημοσιονομικών πλαισίων, δηλαδή μέχρι το 14 και 14 με 20. Ελπίζουμε η έκθεση να αποδώσει. Ε, ειδικότερα ε, θα πρέπει να υπερασπιστούμε αυτή την πολιτική, τη δημοσιονομική, οπότε θα υπάρξει μια έκθεση από την πλευρά ε, δηλαδή, ναι, πράγματι ήταν καλά τα όσα κάναμε γιατί βοηθήθηκε η Ελλάδα. Τώρα, την περασμένη Δευτέρα υπήρξε ε, μια κοινή ε, συνεδρίαση με την Επιτροπή Προϋπολογισμών για τους ελέγχους και εκείνη είχε συντάξει τη σχετική έκθεση για την Ελλάδα το Μάιο του 2017, την οποία όμως εγώ έλαβα μόνο δύο μέρες πριν τη συνεδρίαση. Ε, και ακόμα χειρότερα είναι το, ε, το γεγονός, ή ε, ακόμα χειρότερο είναι το γεγονός ότι ήταν διαθέσιμο μόνο στην ελληνική γλώσσα αυτή η έκθεση. Και εγώ δεν γνωρίζω ελληνικά. Και βέβαια αυτό είναι λυπηρό. Παρ' όλα αυτά όμως θα ήθελα να θέσω έξι ερωτήματα. Ή έθεσα έξι ερωτήματα στον κύριο Παπαστόφ και δεν έλαβα καμία απάντηση στα έξι ερωτήματα που έθεσα και αυτό επιβεβαιώθηκε και από τον Πρόεδρο. Οπότε ε, αυτό με οδηγεί σε μια, ένα συμπέρασμα και ένα ερώτημα από την άλλη πλευρά. Ένα ερώτημα το οποίο ενδεχομένω ε, θα ε, χρειαστεί να αναφέρω και σε μια ολομέλεια γιατί αν δεν λάβω μια απάντηση δεν μπορώ να ε, τοποθετηθώ και στη δική μου έκθεση ως προς το τι τελικά ακριβώς είναι καλό. Άρα λοιπόν ε, θα μπορούσα να λάβω αυτή την έκθεση της ελληνικής κυβέρνησης ε, ε, σε, στη γαλλική, τη γερμανική, την αγγλική, την ολλανδική γλώσσα και όχι στην ελληνική, έτσι ώστε να είμαι σε θέση να την αναγνώσω και να μπορέσω να συντάξω και όπως πρέπει την έκθεσή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαδάκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πριν τις καταστροφικές πλημμύρες στη Δυτική Αττική, ε, οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας είχαν καταθέσει ένα σχέδιο ψηφίσματος στην Επιτροπή Ρέτζη βάζοντας δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτον, το ζήτημα ότι πρέπει το Ταμείο Αλληλεγγύης να αποζημιώνει πληγέντες, δηλαδή εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, και δεύτερον να αρθεί ο απαράδεκτος όρος του 1,5% του ΑΕΠ της Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο ταμείο. Ε, αυτό το ψήφισμα ακόμα είναι στα συρτάρια. Δεν έχουμε ακούσει κάτι. Η κυρία Πρόεδρος ενημέρωσε για οτιδήποτε άλλο μέχρι και για Χριστουγεννιάτικο πάρτι εκτός από αυτό το άμεσο ζήτημα. Συγγνώμη που χαλάμε το χριστουγεννιάτικο κλίμα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν μέσα στις λάσπες αυτή την περίοδο. Και ακριβώς επειδή δεν είναι μία φορά τα 50 χρόνια που έλεγε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο που συμβαίνουν τέτοιες καταστροφές. Πριν από τη Δυτική Αττική ήταν στην ΣΥΜΗ, στην Πιερία, στον Εύρο και μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα έγινε αντίστοιχη καταστροφή και βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι πόλεις της Δυτικής Ελλάδας του Αγρινίου και του Μεσολογγίου. Άρα λοιπόν εξελίσσεται σε πολύ τακτικό φαινόμενο να έχουμε τέτοιες καταστροφικές πλημμύρες που να ε, χτυπιούνται ιδιαίτερα τα φτωχά στρώματα. Κυρία Κρέτσου, ρωτάμε το εξής και ξεκάθαρα. Αναγνωρίζετε ότι πρέπει να έρθουν αυτοί οι απαράδεκτοι όροι του Ταμείου Αλληλεγγύης. Και δεύτερον, τι απαντάτε σε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν με τις λάσπες αυτή την περίοδο το ίδιο πράγμα που απαντήσατε και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λέγοντας ότι περιμένετε το 2020 να συζητήσουμε την αλλαγή των κανονισμών. Γιατί διαφορετικά αυτό συνιστά πολιτικό κινησμό και τίποτα άλλο. Thank you very much. As there was... Ευχαριστώ. Καθώς μου θέσατε ένα ερώτημα θα πρέπει να σας απαντήσω. Ναι, λάβαμε την πρόταση ψηφίσματος στην ελληνική γλώσσα και θα πρέπει να μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης και στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερωθούν οι συντονιστές με βάση δηλαδή τις προβλεπόμενες ε, διαδικασίες ε, του Κοινοβουλίου. Αυτό σε ό,τι αφορά την πρόταση ψηφίσματος ε, στην οποία αναφερθήκατε. Τώρα, ο κύριος Μπούντα είναι ο τελευταίος μας ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκα στο Κλούς με χίλιους ε, δημάρχους και είδαμε τι σημαίνει η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Ξέρουμε ότι είμαστε πολύ ελληματικοί πέρα από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που τόνισε και ο κύριος Μίτελμπουργκ, υπάρχουν και πτυχές που μας οδηγούν στην μη απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Το ΣΥΓΚΕΤ αν και έχει 300.000 κατοίκους, δεν μπόρεσε να εξυγχρονίσει το νοσοκομείο της. Και εγώ ήρθα σε επαφή με επιχειρήσεις για να δούμε γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτός ο εξυγχρονισμός και δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορούσαν να απορροφηθούν τα κονδύλια. Υπάρχουν οικονομικοί πόροι για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Υπάρχουν όμως και ερεσιμότητες. Δηλαδή ότι αυτά τα κτίρια θα πρέπει να συνδέονται με το κεντρικό δίκτυο θέρμανσης. Μα εμείς είμαστε μια αγροτική περιοχή, δεν μπορούμε να συνδεθούμε με το κεντρικό δίκτυο. Και μέσα στα πλαίσια και αυτής της Επιτροπής αλλά και της Άγκρη μιλήσαμε για την απερίμωση αυτών των περιοχών. Και είναι δύσκολο να υπάρχει σωστή υδροδότηση αυτών των περιοχών. Δυστυχώς όμως υπάρχει και εκεί ε, αιρεσιμότητα, ότι δηλαδή ε, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες περιφέρειες που να υπερβαίνουν τους 2.500 ε, κατοίκους. Εμείς ξέρετε ότι δεν έχουμε κάνει απογραφή εδώ και πολλά χρόνια και δεν μπορούμε να δώσουμε τα μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους για να μην εγκαταλείψουν αυτές τις περιφέρειες. Δηλαδή αυτά τα χρήματα αν και τα διαθέτουμε στους πολίτες, δυστυχώς ε, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από περιφέρειες οι οποίες έχουν απεριμωθεί. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές που να ζητούν το λόγο, επιτρέψτε μου να θέσω ένα ερώτημα και από τη μου πλευρά. Εγώ δηλαδή, ως ε, πρόεδρος. Και αυτό το ερώτημα προέκυψε μετά από τη συζήτηση που άκουσα εδώ στην Επιτροπή ΡΕΙΤ. Μας είπατε, Επιτροπή, ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η έκθεση εφαρμογής. και βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει κατά τι τελευταίε εβδομάδε μία σειρά από διαφορετικέ πρωτοβουλίε από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να διαμορφώσουμε τη δική μας ε, θέση ως ε, Επιτροπή Ρέτη και ως ε, Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την 7η έκθεση συνοχής ακριβώς για την χάραξη της μελλοντική πολιτικής συνοχής μετά το 2020. Έχουμε συμμετάσχει σε διαφορετικές εκδηλώσεις, σε διαφορετικά επίπεδα και εκεί έχουμε λάβει πολύ σημαντικά μηνύματα ε, σε ό,τι αφορά τις ε, περιφερειακές ε, πολιτικές, σε ό,τι αφορά τις, τα κονδύλια και την ανάγκη δηλαδή χρηματοδότησης και βέβαια αυτή η ανάγκη μπορεί να καλυφθεί μόνο από τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής. Και εδώ έρχομαι στο, στα όσα είπε ο συνάδελφος Νοβάκο. Δηλαδή, από τώρα μέχρι την έναρξη του επόμενου πολιτού σε δημοσιονομικού πλαισίου έχετε προβλέψει κάποια χρηματοδότηση και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς από την πλευρά μας για να υποστηρίξουμε ε, αυτή την κοινή προσπάθεια για τη χάραξη της μελλοντικής πολιτικής συνοχής. Ε, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι υπάρχει υποστήριξη από την πλευρά του Συμβουλίου, αλλά γνωρίζουμε ότι στο Συμβούλιο υπάρχουν μια σειρά από διαφορετικά συμφέροντα που πρεσβεύουν τα διαφορετικά κράτη-μέλη. Οπότε εμεί από την πλευρά μα ναι υποστηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία, είμαστε διατεθειμένοι να εργαστούμε περαιτέρω επ' αυτού και θα συζητήσουμε μάλιστα και τα επόμενα βήματα στην συνεδρία των συντονιστών που θα έχουμε σήμερα. Αλλά εσεί από την πλευρά σα, Επίτροπε, τι έχετε να μα πείτε σε σχέση με αυτό. Αυτό ήταν το ερώτημά μου και δίνω ε, το λόγο σε εσά, κύριε Επίτροπε. Thank Ε, σας ευχαριστώ πολύ. για όλα αυτά τα διαφορετικά ερωτήματα που μου θέσατε. Συμμερίζομαι κάποιες από τις ανησυχίες σας και όπως είπα και κατά την αρχική μου παρέμβαση, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία πριν από το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και θα ξεκινήσω εδώ από αυτό που είπε η πρόεδρος μόλις τώρα, ότι θα πρέπει να γίνει μια κοινή προσπάθεια, ας μην πω κοινό αγώνας ε, εκείνη μάχη μπροστά μας. Δεν είναι τόσο διπλωματική αυτή η έκφραση. Ε, άρα λοιπόν μια κοινή προσπάθεια αποκινούμε όλου του όλους τους συναρμόδιους φορείς προκειμένου να προωθήσουμε τα στοιχεία εκείνα που είναι θετικά, ε, την πολιτική δηλαδή η οποία είναι πιο εφικτή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η πολιτική συνοχής να διατηρηθεί. Τώρα, θα απαντήσω στα ερωτήματα με τη σειρά που τέθηκαν. Ε, αρχικά να πω, να χαιρετήσω εδώ τους ε, επισκέπτες μας ε, που έχουμε από το Σαν Μάρτιν και το Σαν Μαρτέν. Δεν ξέρω πώς προφέρεται ακριβώς η Ολλανδική πλευρά, το Μάρτιν. Πάντως, εγώ είχα τη δυνατότητα να συναντήσω τον πρόεδρο της γαλλικής πλευράς όταν είχα επισκεφθεί τη Γαλλική Γουιάννα γιατί είχε αναλάβει η Γαλλική Γουιάννα την ε, Προεδρία των πλέον απομακρυσμένων περιοχών, οπότε είχα ε, τη δυνατότητα εκεί να επισκεφθώ τον Πρόεδρο του Διαμαρτίου, να αποκοινούμε τον ε, Πρόεδρο Μακρόν και σε αυτό το πλαίσιο δημοσιεύθηκε και ανακοίνωση τη Επιτροπή σε ό,τι αφορά τι πλέον απομακρυσμένε περιοχέ και ο εισηγητή ήταν ο κ. Ματσού, ο οποίο δεν παρευρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ, αλλά ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Κάθε μέρα μαθαίνουμε κάτι καινούριο και εκείνο που μπορώ να σα πω είναι ότι για μένα αποτέλεσε έκπληξη όταν είδα για πρώτη φορά το σχετικό φάκελο ότι η Ολλανδική πλευρά του Αγίου Μαρτίνου ουσιαστικά δεν θεωρείται τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτό δηλαδή δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην υποστήριξη αυτής της πλευράς. Αλλά από την πρώτη στιγμή βέβαια υπήρξε αλληλεγγύη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αξιοποιήσαμε όλα, ενεργοποιήσαμε όλα τα, ε, τις δυνατότητες, τους μηχανισμούς παροχής έκτακτης βοήθειας που είχαμε στη διάθεσή μας και υποστηρίξαμε και τις κάτω για την υποστήριξή τους απέναντι στον Αγιο Μαρτίνο και μέσω παροχής δορυφορικών υπηρεσιών ε, κατά την πρώτη εβδομάδα μετά την καταστροφή αλλά και κάτι γενικότερο περίοδο της κρίσης. Ε, γνωρίζω δηλαδή πως ο πρόεδρος Γιούνκερ ε, συνομίλησε και με τον ε, Πρωθυπουργό των Κάτω Χωρών ως το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και επίσης ο μηχανισμός ανταπόκρισης, αντιμετώπισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν συνεχώς διαθέσιμος, σε επαφή δηλαδή με όλους τους συνθήνοντες σε αυτή την περιοχή, ειδικότερα την Ολλανδική πλευρά. Επίσης ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ήδη χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα Interreg ε, για την ανακατασκευή των ε, υποδομών και στις δύο πλευρές, δηλαδή και στο γαλλικό και στο ολλανδικό τμήμα. το Ολλανδικό δηλαδή ε, τμήμα του νησιού σε ό,τι αφορά αυτή την, την αναποκατάσταση των υποδομών μπορεί να καλυφθεί ε, έως και κατά 3 εκατομμύρια ευρώ. Ε, τώρα, ε, στην προηγούμενη εβδομάδα στη διάσκεψη κορυφή σε ό,τι αφορά την Καραϊβική, ο κύριος Μίτσα ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν άλλα 300 εκατομμύρια ευρώ σαν αναπτυξιακή βοήθεια στις, ε, στην περιοχή της Καραϊβικής. Ε, σε συνέχεια βέβαια ακριβώς των πρόσφατων καταστροφών των τελευταίων κυκλώνων Ήρμα και Μαρία. Νομίζω πως θα ήταν μια καλή ιδέα να υπάρξει εδώ ένας συντονιστής για αυτό το ζήτημα και θα έρθω σε επαφή με τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους και τις υπηρεσίες της Επιτροπής για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί έχετε ε, δίκιο όταν λέτε ότι έχουμε διαφορετικά εργαλεία, δηλαδή το Interreg που ανοίγει στη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο, μετά έχουμε το άλλο εργαλείο που ανήκει στην ΤΕΦΚΟ, οπότε θα μπορούσαμε ενδεχομένω να δημιουργήσουμε μια ομάδα εργασία η οποία θα βρίσκεται σε επαφή τόσο με το Ολλανδικό όσο και το Γαλλικό Τμήμα του νησιού. Πάντως ε, πραγματικά συμφωνώ μαζί σας ότι χρειαζόμαστε μία ενοποιημένη, μία ολοκληρωμένη προσέγγιση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, αποκατάσταση και των δύο πλευρών του νησιού και νομίζω ε, πως ε, οι τοπικές αρχές και των δύο πλευρών του νησιού θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια ευρύτερη συνεργασία ανάμεσα στις αρχές των δύο πλευρών του νησιού από την πλευρά τη Επιτροπή, εγώ σα διαβεβαιώ ότι θα κάνουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει συμπληρωματικότητα ανάμεσα στι παρεμβάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και ε, τι παρεμβάσει και τα έργα τα οποία ε, τρέχουν σε τοπικό επίπεδο. Και επίσης ε, θα δούμε πώς ε, στο πλαίσιο των μελλοντικών ε, προγραμμάτων μπορούμε να έχουμε καλύτερη ε, στόχευση για την αποκατάσταση των αποδομών σε συνέχεια των δικλώνων Ήρμα και Μαρία. Πραγματικά ε, έχουμε λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτές τις καταστροφές. Δεν έχω συναντηθεί κομματιμερός με τους δύο εκπροσώπους, αλλά μπορούμε να το κάνουμε στη συνέχεια εδώ της συνεδρίασης για 10 λεπτά. Ε, και ε, σας είπα ότι συνομίλησα με τον πρόεδρο Γιούνκερ για αυτό το ζήτημα και στο πλαίσιο της Γαλλικής Γκουιάνα και επίσης συνομίλησα με τον πρόεδρο του Γαλλικού Τμήματος. Υπάρχουν και κάποια κονδύλια στο πλαίσιο του ERDF, δηλαδή του Ταμείου Περιφερειακής ανάπτυξη, τα οποία θα μπορούσαν και αυτά να αξιοποιηθούν για την αλκοδόμηση. Οπότε πραγματικά σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει αλληλεγγύη από την πλευρά μας και ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να ε, βοηθήσουμε εσάς, αλλά και βέβαια με την ταυτόχρονη βοήθεια των εμπλεκόμενων κρατών μελών, δηλαδή της Γαλλίας και των ε, κάτω χωρών. Και από εκεί και μετά θα λάβουμε υπόψη μας και την πρόταση συντονισμού στην οποία αναφερθήκατε τώρα. Σε ό,τι αφορά την Οικονομική και Νομισματική Ένωση του ΕΜΙΟ, κάτι το οποίο έθεσε και ο κύριος Βανίστελρο, αλλά και η κυρία Κρέλ, όπως ανέφερα προηγουμένως, ένα συγκεκριμένο, ένα ιδιαίτερο ζήτημα του χθεσινού πακέτου αφορά την πολιτική συνοχή και μάλιστα είναι σημαντικό το ζήτημα αυτό και αφορούσε την πρόταση για την τροποποίηση ε, του CPR, δηλαδή του κανονισμού για τους γενικούς ε, κανόνες και του σχετικού αποθεματικού ε, και εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι αυτή η δυνατότητα θα είναι εθελοντική. Οπότε, τώρα, η πρόταση έγινε από την πλευρά της Επιτροπής και εμείς από την πλευρά μας τώρα αναμένουμε τον επικοδομητικό διάλογο που θα ακολουθήσει με την Επιτροπή ως συνομοθέτη. Τώρα, απαντήσω στον κύριο Τόμασίτς. σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα πολυταμιακή χρηματοδότηση στο πλαίσιο τη ε, μελλοντική νομοθεσία. Νομίζω πω είναι πολύ σημαντικό το σχόλιο που κάνατε. Δηλαδή, υπάρχουν τόσο καλά, πολλά καλά παραδείγματα, τα οποία θα πρέπει να αναδείξουμε περαιτέρω, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε πράγματι να επιτύχουμε περισσότερε ε, συνέργειε ε, στο πλαίσιο τη ε, επόμενη για παράδειγμα, πρόταση που θα κάνουμε. Να είναι δηλαδή δυνατό να ε, αξιοποιούνται τις συνέργειες ευκολότερα. Και νομίζω πως ε, είναι σημαντικό αυτό και στο πλαίσιο τη της πρότασης του κανονισμού Omnibus ε, που βρίσκεται στην τελευταία φάση. Δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε ένα ακόμα τριμερή διάλογο και ελπίζουμε εκεί να καταλήξουμε. Εκεί λοιπόν θέλουμε ακριβώς να προβλέψουμε τη διευκόλυνση της, του συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών χρηματοδοτήσεων των διαφορετικών ταμείων. Έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει συγχρηματοδότηση από τα ταμεία. Ε, τώρα σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα, τα financial instruments, ε, ναι, πράγματι έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε ότι έχουν ξεκινήσει καθυστερημένα τα κράτη-μέλη να τα αξιοποιούν και στην ε, ε, περίοδο 2017-2013 αυξήθηκε, 2007-2013 αυξήθηκε η αξιοποίησή τους και τώρα θέλουμε Ε, και βλέπουμε οτι περισσότερη αξιοποίηση. Υπάρχουν μόνο δύο κράτη-μέλη τα οποία πραγματικά δείχνουν να είναι ακόμα επιφυλακτικά απέναντι σε αυτή τη χρηματοδοτική λύση, αλλά προσπαθούμε να τα πείσουμε να αλλάξουν στάση, γιατί κατά τη δική μας άποψη έχει χρησιμότητα. Δηλαδή, για κάθε ένα ευρώ που θα έχει επενδυθεί, στο πλαίσιο της περίοδου 2014-2020, στο πλαίσιο αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων, θα έχουμε 3 ε, έως 4 ε, ε, ευρώ έως το 2023. Και εδώ αναφέρομαι και στο σχέδιο Marshall, το οποίο είχε σχεδιαστεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι υπάρχουν δύο χώρε, η Αυστρία και η Γερμανία, που ακόμα επαναχρησιμοποιούν, ανακυκλώνουν, αν θέλετε, αυτά τα κονδύλια που είχαν λάβει από το σχέδιο Μάρσαλ. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι απλώ μια θεωρία. Είναι κάτι το απτό, κάτι το πραγματικό. Είναι δυνατό να αναχρησιμοποιεί, να επαναχρησιμοποιεί κανεί τέτοια κονδύλια. Δηλαδή μπορεί κανεί να επενδύει ένα ευρώ και τελικά να μένουν στα χέρια του πέντε ευρώ από την επένδυση που έχει κάνει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τα κράτη-μέλη απέναντι σε αυτή τη δυνατότητα και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Αλλά για να το επιτυγχάνουμε χρειαζόμαστε και τεχνογνωσία αλλά και την κατάλληλη διοικητική ικανότητα. Εσεί ε, προέρχεστε από την, κατάγεστε από την Κροατία, έτσι. Ναι, ε, από τα συστήματα μπάνξης έχουμε δει κάποιους υπουργούς πάρα πολύ ε, καλού και οι οποίοι γνωρίζουν πώς μπορούν να τα, τα σχετικά συστήματα. Και νομίζω δηλαδή πως οι υπουργοί σας ε, γνωρίζουν καλά πώς ε, μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την καλύτερη εφαρμογή, ε, νομίζω πως εδώ η δουλειά θα ξεκινήσει από κοινού. Η συζήτηση δηλαδή θα ξεκινήσει αμέσως μετά το ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο δηλαδή θα υποβληθεί τον Μάιο του 2018. Οπότε λοιπόν το συντομότερο δυνατό μετά από τον Μάιο του 2018 θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τη νέα νομοθεσία και τους τρόπους που μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Εκείνο όμως που μπορώ να σας πω είναι πως εφόσον θα πληρούνται οι προτέρων ερεσιμότητες ε, για αυτή την περίοδο σε πολλές ε, περιοχές δεν θα είναι απαραίτητο πλέον να εφαρμόζονται. Δηλαδή ναι, χάσαμε λίγο χρόνο αυτή την περίοδο, αλλά αυτό ήταν καλό. Γιατί διάφορα κράτη-μέλη δεν θα είχαν εστιάσει στρατηγικές του, για παράδειγμα, στην ίδρυψη, στην υγεία, στις μεταφορέ ή οπουδήποτε αλλού, χωρί να υπάρχουν οι εν λόγω εκ των προτεραιών αιρεσιμότητε. Και εφόσον θα έχουν εκπληρωθεί για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, δεν θα χρειάζεται κατά την έναρξη τη επόμενη προγραμματική περίοδου να σπαταλήσουν τόσο χρόνο σε αυτές τις ίδιες ερεσιμότητες. Οπότε θεωρώ πως ήταν πολύ καλή ιδέα αυτέ οι ερεσιμότητε και θα, είναι, θα έχουν μεγάλο βάθο χρόνου, δηλαδή θα προκύπτουν ξανά και ξανά κατά την έναρξη κάθε προγραμματική περίοδου, όχι, απλώ θα παρακολουθούνται ω προ το αν συνεχίζουν να πληρούνται ή όχι εν λόγω ερεσιμότητες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημα ε, που έθεσε ο κύριος Βαν Μίλτεμπουργκ ε, αναφέρθηκα ήδη στο ζήτημα της Οικονομικής Ένωσης και στο ζήτημα του Αγίου Μαρτίνου, αλλά όπως είπα θα διαβιβάσω στους συναδέλφους της Επιτροπής ε, την πρόταση που κάνατε. Τώρα, ένας χρηματοδοτικός συντονισμός ίσως θα πρέπει να υπάρξει ανάμεσα στον εθνικό συντονισμό στη Γαλλία, τον εθνικό συντονισμό στις κάτω χώρες και τον συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας ε, είπα ε, ποια είναι περίπου τα κονδύλια τα οποία έχει ε, ανακοίνωσε ο κ. Μίμετς πως έχουν ήδη δεσμευτεί για χρηματοδότηση στην περιοχή της Καραβικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Ρουμανία. Αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω, θα μιλήσω στη μου γλώσσα. Uh... Γνωρίζετε πολύ καλά πώς έχει κατάσταση. ευχαριστώ για την παρουσία σας στο Κλούζ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ τον κύριο Μπούντα για την οργάνωση. Ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η επίσκεψη. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά τη Ρουμανία όπως και όλα τα άλλα κράτη-μέλη καταρχήν την κυβέρνηση και τις ε, εθνικές αρχές, οι οποίες ε, είναι απαραίτητες για να αξιοποιηθεί 100% αυτή η βοήθεια. Για την περίοδο 7-13 οι υπηρεσίες μας κάνανε ό,τι μπορούσαν για να υπάρξει σωστή απορρόφηση ε, δυστυχώς δεν υπήρχε απόλυτη επιτυχία, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών. Ιδιαίτερα για τα σχέδια που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015. Θα χρησιμοποιηθούν ακόμα τα χρήματα που ισχύουν για το πολιετές 14-20 τα νέα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ρουμανία, θα πρέπει να θεωρήσουν την πολιτική συνοχής ως μια μεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Όπως ξέρετε, ε, μεταξύ 2007 και 2013 υπήρξε απορρόφηση της τάξης του 89 μέχρι 91%. Στον τομέα των ε, μεταφορών είναι ελληματική. Ως προς την τρέχουσα ε, χρηματοοικονομική διαδικασία, όχι μόνο στη Ρουμανία υπάρχει χαμηλότερος ρυθμός απορρόφησης κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι προσπάθειες έτσι ώστε η Ρουμανία να μπορέσει να αδράξει την ευκαιρία που τις προβάλλεται τη στιγμή που έχει και έναν από, το, τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρες της πρώην ε, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Δυστυχώς η πολιτική αστάθεια είναι ένας αρνητικός παράγων. Ε, εγώ τρία χρόνια διανύω σε αυτή μου τη θέση και ήδη διαπραγματεύω με το τέταρτο πολιτικό σχήμα που δημιουργήθηκε. Το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα αυτό. Όμως ε, υπάρχει καλύτερη διαχείριση. Έχουμε λάβει τις πρώτες ε, αποδείξεις και μεγάλες συμβάσεις που θα ε, θα γίνουν πάρα πολύ μεγάλες μάλλον απορροφήσεις από, αυτά τα, ε, από τις μεγάλες συμβάσεις οι οποίες μας απεστάλησαν. Στις 18 και 19 Δεκεμβρίου θα ε, επισκεφθώ εκ νέου στην Ρουμανία. Συμφωνώ μαζί σας. Ήρθα σε επαφή με τους ε, δημάρχους, η πόρτα είναι ανοιχτή, όπως και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Ρότερταμ συναντηθήκαμε με 600 δημάρχους και με βάση αυτή την αστική ατζέντα για πρώτη φορά οι πόλεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Και 1,2 δις, δηλαδή 20% των πόρων, την χάνουν ε, διαχείρισης ε, από τις πόλεις. Θα έρθω σε επαφή με τις ε, υπηρεσίες μου. Ξέρετε, ότι υπάρχει 1,5 ε, δις για την υποστήριξη των νοσοκομείων, μεταξύ των οποίων και του νοσοκομείου του ΣΥΓΚΕΤ. Δυστυχώς στη Ρουμανία ε, δεν εργαζόμαστε όπως ε, στη Γερμανία για παράδειγμα όπου κάθε περιφέρεια είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των πόρων της. Δεν υπάρχει αυτή η αυτονομία, η διοικητική αυτονομία. Νομίζω ότι η παρούσα ε, διαχείριση δυσχεραίνει τα πράγματα γιατί παρά τις ε, δυσκολίες βρισκόμαστε σε μια κατάσταση βελτίωσης με την ε, συνεργασία των ε, νομαρχιακών και τοπικών αρχών και αυτές τις μέρες μια ομάδα εμπειρογδομόνων της Επιτροπής και της Παγκόσμιας Τράπεζας βρίσκονται στην Πιάτρα Νεάμτς για να δούμε την διαδικασία επιλεξιμότητας των περιφερειών. Είχαμε ένα εκατομμύριο που δώσαμε στην Πολωνία για αυτόν τον πυλώνα και για τη Ρουμανία φτάσαμε σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο και δώσαμε ακόμα 500.000, δηλαδή 1,5 σύνολο εκατομμύριο όπως συμφωνήσαμε με την κυρία Ροβάνα Πλούμπ. Πρόκειται για μια εταιρική σχέση η οποία είναι πρωτόγνωρη μέσα στα πλαίσια της ε, διαχείρισης των πόρων μεταξύ περιφερειών του ε, Βορρά και του Νότου ως προς την ενεργειακή απόδοση θα ήθελα να σας πω ότι δεν υπάρχει αυτός ο όρος του ελάχιστου παρονομαστή κατήχων 2.500. Κύριε Μπούντα, βρέθηκα στο κλούς και θα ήθελα να πω ότι μετά από 10 λεπτά χαλαζόπτωση ε, δεν είχα ούτε ηλεκτρικό ούτε νερό. Σας μιλώ για τη δική μου επαρχία που είναι ακριβώς έξω από το κλούς. Δηλαδή με σταματούσαν άνθρωποι στους δρόμους και μου λέγαν σας παρακαλώ ε, μιλήστε για το δίκτυο ίδρευσης. Είναι απαράδεκτο τον 21ο αιώνα να μην λειτουργούν σωστά, να μην ε, λειτουργεί το δίκτυο ίδρευσης και να μην έχουμε δυστυχώς νερό καλής ε, ποιότητας στη Ρουμανία. Ξέρετε πόσοι ε, νέοι εγκαταλείπουν την ύπεθρο, δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 75 χρόνια σε πολλά χωριά της ε, Ρουμανίας και όχι και ιδιαίτερα απομακρυσμένα. Συζητήσαμε με τις τοπικές αρχές, αλλά όλα εξαρτώνται και από τους δημάρχους. Συμφωνώ ότι κάτι θα πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να ανακτήσουν ε, πληθυσμό αυτές οι περιφέρειες. Μιλάμε για αστική ατζέντα χωρίς την κατάλληλη ε, υποδομή. Έχουμε μεγάλα άστεα που συγκεντρώνουν το 80% του πληθυσμού, αλλά δεν μπορούμε να ε, μεταφέρουμε τον πληθυσμό μακριά από τα αστικά κέντρα. Αυτό το συζητήσαμε και με τον Επίτροπο Χόγκαν. Θα πρέπει να βοηθήσουμε όχι μόνο τους ε, αγρότες, αλλά και τους ε, πολίτες που δεν πρέπει να απομακρύνονται από τη γενέτειρά τους. Κύριε Χόπ, εδώ και έξι χρόνια έχουμε στη διάθεσή μας αυτό το μέσο, δηλαδή νήσιν 3. Άρα μπορεί να εφαρμοστεί ε, μέχρι ε, το 2023. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, πλουστευμένους μηχανισμούς, μιλήσατε για εξάντε ερεσιμότητα και φυσικά δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο για τη μελλοντική περίοδο. Και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα καταφέρει να εγκρίνει τη νομοθεσία για μετά το 2020 για να μην έχουμε καθυστερήσεις. Κυρία Μάτο, ξέρετε... Ξέρετε ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι στο επίκεντρο της πολιτικής. Είναι κάτωθεν προσέγγιση που βασίζεται στην τοπική αυτοδίκηση. Πρόθεσή μου είναι να συνεργαστώ μαζί σας. Γνωρίζω ότι στην Ιταλία, όπως και σε άλλα κράτη-μέλη, όπως σας είπα, δεν αποτελεί παράδοση όπως στην Ολλανδία και όπως σε άλλες χώρες να λαμβάνονται υπόψη όλες οι θέσεις, αλλά ελπίζω πραγματικά ότι οι Ιταλικές αρχές κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να διαμορφώσουν καλές στατικές της περιφερής. Για το Ταμείο Λιλεγγύης γνωρίζω πολύ καλά όλες τις απογοητεύσεις που έχουμε όλοι μας όταν δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Θα επανέλθω σε αυτό όταν θα απαντήσω στον κύριο Παπαδάκη για το θέμα αυτό. Κυρία Νταμάτο, να σας πω ότι η νέα πρόταση για ίσως να είναι καλύτερη για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να επανεξετάσουμε τις συνθήκες χρήσεως του Ταμείου Αλληλεγγύης. Δεν είπα στην Ολομέλεια, κύριε Παπαδάκη, ότι πρέπει να περιμένουμε το 2020. Σας σέβομαι πάρα πολύ, αλλά σας λέω ότι νομίζω ότι ήταν άδικο αυτό να πείτε ότι είμαι κοινική γι' αυτό. Δέκα φορές ήρθα, εννέα φορές ήρθα εδώ σε εσά. Άλλαξα τον κανονισμό, ήταν εξαιρετη, έκτακτη αλλαγή του κανονισμού για την Ελλάδα. Μοιράζομαι ποιο στην άποψή σα. Μίλησα με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, την Παρασκευή για τι πλημμύρε. Το εξήγησα και του είπα ότι τον Απρίλιο-Μάη θα αλλάξει η νομοθεσία και το 2020. Το κανονισμό, συγγνώμη. Θα αλλάξει ο προπολογισμό τον Μάη αμέσω μετά την αλλαγή της νομοθεσίας και του κανονισμού. Και όλα αυτά τα όρια υπάρχουν και προβλέπονται και οι προϋποθέσεις λόγω του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τα υιοθέτησαν. Δεν ήταν έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το όριο. Κατανοώ, καταλαβαίνω τα τεράστια προβλήματα που έχουμε στην Αττική, αλλά σύμφωνα με τον κανονισμό που υιοθετήσατε, η Αττική είναι η πλουσιότερη περιοχή περιφέρεια. Και οι προσπάθειες ευρωπαϊκέ πρέπει να συνάδουν με τις ελληνικές προσπάθειες, να πηγαίνουν χέρι με χέρι οι προσπάθειες αυτές. Συγγνώμη σας το λέω, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι ήταν άδικο απέναντί μου και απέναντι στις υπηρεσίες μας. Όταν προσπαθούμε να βοηθούμε όσο γίνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε απολευθερώσει τη ρευστότητα, έχουμε μπροστά μας αυτό το κανονισμό το σχετικό, παρά, πολεμούμε παρά τον δισταγμό των 100 μελών για την Ελλάδα να κάνουμε 100% χρηματοδότηση, από, ξεμπλοκάραμε όλα τα προγράμματα, ξεκινάμε, εγγενιάσαμε το τέμπι. Έχουμε ξεκινήσει, εγγενιάζουμε και τα έργα για το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Καθημερινά εργαζόμαστε στην Ελλάδα για αυτό το θέμα και φυσικές καταστροφές είναι συμβάντα που συμβαίνουν όλο και πιο συχνά. Εγώ είμαι υπέρ των να επεξετάσουμε, αλλά δεν γίνεται, δεν πρέπει τον κανονισμό να γίνεται μία νυχτή από τη μία μέρα στην άλλη. Ήμουν στην Πορτογαλία, μόλι ήρθα από την Πορτογαλία. Είδα τι καταστροφέ, τι πυρκαγιέ, στη Μαδέρα επίση, στην Ελλάδα. Μη λέτε λοιπόν ότι δεν δείχνουμε αλληλεγγύη, δεν μπορείτε να το λέτε αυτό. Πανεξετάζουμε τον κανονισμό για την πολιτική προστασία. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε να γινόμεθα πάρα πολύ πιο γρήγορα, να είμαστε πιο ευέλικτοι. Επίσης όμως θα πρέπει να συνεργαστούμε χέρι με χέρι με τα κράτη-μέλη και εκφράζω για μία ακόμη φορά τα συλληπιτήριά μου για αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα και προσπαθούμε με τον Υπουργό τον αρμόδιο, μίλησα και με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργό, ο κύριο Τσίπρα, μίλησε με τον πρόεδρο Γιούνκερ. Προσπαθούμε να εξετάσουμε τον κανονισμό από κάθε οπτική γωνιά, να δούμε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε. Θα βοηθήσουμε την Ελλάδα. Μέχρι τέλους, όσο μπορούμε, να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα έχει ένα πόρο που έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. 1,3 δισεκατομμύρια σε αυτή την προγραμματική περίοδο για την πρόληψη του κινδύνου και αλλαγή του κλίματος. Και η Ελλάδα αν είχε έργα, προγράμματα, μπορούσε να χρησιμοποιήσει περισσότερα από τα χρήματα. Τα χρήματα υπάρχουν. Έχουν διατεθεί για την Ελλάδα. Δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα καλών προγραμμάτων, ε, προλήψεως των κινδύνων και νομίζω ότι κάναμε πολλά. Βέβαια υπήρξαν πολλές καταστροφές. Ταυτόχρονα όμως με το μηχανισμό προλήψης του κινδύνου και που σπρώξαμε την Ελλάδα να έχει ε, ειδική στρατηγική, έχουμε αποφύγει πολλές ακόμα ανθρώπινες τραγωδίες. Βέβαια, είναι μια τραγωδία αυτή που συνέβη για όλους μας. Αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα, αυτά που συμβαίνουν στην Πορτογαλία, όλους μας πλήττουν. Ε, ε μας πληγώνουν θέλω να πω. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε, σε διαβεβαιώνω. Από τον Ιούνιο ήδη θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να επαναξετάσουμε τους όρους για τη χρήση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι καλή στιγμή να κάνουμε ε, μια αποτίμηση και να δούμε πώς αυτό το Ταμείο Αλληλεγγύης μπορεί να αλλάξει υπέρ κάποιων κρατών μελών. Στον κύριο Μπούντα απάντησα για την εφαρμογή και την υλοποίηση τώρα. Όπως σας είπα, τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η εκτέλεση έχει φτάσει τον κανονικό ρυθμό. Είμαστε κοντά στο μισό των διαθέσιμων πόρων για το 2014-2020 που έχουν ε, δεσμευτεί για τα προγράμματα. Αυτό συνάδει με το ρυθμό εφαρμογής περίοδο 2007-2014. Ε, Όπως σα είπα, περισσότερε λεπτομέρειες θα είναι διαθέσιμε στην έκθεση που θα υιοθετηθεί στις 13 ε, Δεκεμβρίου. Να σας πω ότι είμαι εξίσου απογοητευμένη που αυτή η επιλογή των προγραμμάτων δεν αντικατοπτρίζεται στις πληρωμές που κατεβλήθησαν. Συνάντησα τον Υπουργό σας, τον Υπουργό τον Υπουργό Οικονομίας της Ολλανδίας και εξεπλάγει η κυρία αυτή που άκουσα να της λέω ότι περιμένουμε ε, για τις πληρωμές, σχέδια πληρωμών. Ε, έχουμε ε, πολλά χρήματα που θέλουμε να δώσουμε στην Ολλανδία. Ξεκινήσατε με τα δικά σας χρήματα, με τα δημόσια χρήματα, ίσως και ιδιωτικά χρήματα και δεν έχουμε λάβει τις αξιώσεις για, τι για Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. Π.χ. ότι εμείς ήδη έχουμε ε, εργαστεί επί τόπου, έχουμε κάνει την προετοιμασία και περιμένουμε ε, για, τις, ε, για τα τιμολόγια. Βέβαια, συμφωνώ μαζί σας ότι η έναρξη της εφαρμογής ήταν καθυστερημένη, ήταν αργή, μη ότι όλη η νομοθεσία υιοθετήθηκε εδώ στο Κοινοβούλιο αρκετά αργά για το 2014-2020 και χρειαζόμασταν κάποιο χρόνο ούτως ώστε οι αρχές να αντιμετωπίσουν τις καινοτομίες του, της νέας νομοθεσίας και για την προετοιμασία των διαφόρων προγραμμάτων. Η εκτέλεση αυξήθηκε, ο ρυθμός εκτέλεσης σημαντικά το τελευταίο έτος και φτάνει τους ρυθμούς τους αρχικούς και καλύπτει τις χρονικές καθυστερήσεις. Μιλάμε για 2014-2020 για αυτή την περίοδο, αλλά έχουμε άλλα έξι χρόνια μέχρι το 2023. Ο κύριος Νοβάκοφ. Κύριε Νοβάκοφ, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι απάντησα στον Λάμπερτ και Κωνστάνσε στα μέλη αυτά για το απόθεμα, για τις μελλοντικέ συζητήσεις και τις συνεχιζόμενες. Προσβλέπουμε στη συμβολή της Επιτροπής σας, κυρίως μέσω της εκθέσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 7η ε, Πολιτική Συνοχής. Δεν σας αποκρύπτω ότι βασιζόμαστε πολύ στην κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρο, ε, τον κύριο Νοβάκοφ και τη Βουλγαρική Προεδρία. Τι μπορούμε να κάνουμε, να συνεργαστούμε. Είπε και η κυρία Πρόεδρος. Είναι καλό ότι έχουμε το Συμβούλιο στο πλευρό μας όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων. Να δούμε τι θα γίνει Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Στη Σόφια θα συναντήσει ο κ. Έτιγκερ τον Υπουργό Οικονομικών, μάλλον του Υπουργού Οικονομικών, για το Ταμείο Αλληλεγγύης. Απάντησα σας είπα, βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας η σύσταση του Ταμείου αυτού. Οι συνομοθέτες αποφάσισαν ότι παρεμβαίνει το Ταμείο Λιλεγγύης όταν φτάσει η καταστροφή ε, σε κάποια επίπεδα τέτοια που δεν μπορεί το κάτω μέλος να αντιμετωπίσει την καταστροφή ε, μόνο του. Γι' αυτό τέθησαν για κάθε χώρα κάποια όρια και κάθε περιοχή για την κινητοποίηση του Ταμείου. Όταν εδώ και 1,5 χρόνο δημιουργήθηκε το Ταμείο, συζητήσαμε εκτενώς με τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο αυτά τα όρια κινητοποίηση του Ταμείου. Τον Μάη, όπω σα είπα, μαζί θα πρέπει να το κουβεντιάσουμε το θέμα, διότι αισθάνομαι ότι χρειαζόμαστε περισσότερο περιθώριο ελιγμών. Είναι προφανές αυτό για μένα. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά δεν χρειάζεται να αλληλοκατηγορούμεθα. Είμαστε ο ένα στο πλευρό του άλλου στην πραγματικότητα. Για τα ειδικά μέτρα, για τα συγκεκριμένα μέτρα για την Ελλάδα, διότι α, μιλώσαμε γι' αυτό, σύμφωνα με τις τροπολογίες που αφορούσαν τα ειδικά μέτρα για την Ελλάδα, ξέρετε πολύ καλά ότι οι ελληνικές αρχές και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόνο οι ελληνικές επιτροπές που να την έκθεση για την εφαρμογή των μέτρων οι ελληνικές αρχές συνέταξαν και υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σχετική έκθεση και στην Ελλάδα το έχετε λάβει η μετάφραση εκτελείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας ενημερώσουμε αμέσως ε, αξιότιμε κύριε Βουλευτά γιατί όλοι ενδιαφερόμαστε θέλουμε η Ελλάδα να λύσει τα προβλήματα. Τώρα, ξέρετε ότι στην προηγούμενη περίοδο είχαμε επιλέξει 181 προγράμματα. Τώρα θέλουμε να εστιαστούμε στα σημαντικότερα, στις ανάγκες, στις μεγαλύτερες. Πώς έχουμε? 18 προγράμματα στα οποία επικεντρώνουμε, στο μετρό της Θεσσαλονίκη και άλλα σημαντικά έργα, ούτως ώστε να επιταχυνθεί η εφαρμογή, η εκτέλεση και να δούμε την πρόοδο. Θα είμαστε επαφή μαζί σας και θα έχουμε έτοιμες και τις διάφορες γλωσσικές εκδοχές του κειμένου. Κυρία Μιχαήλοβα, σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Ευχαριστώ όλα τα μέλη, όλες τις πολιτικές ομάδες κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. Οι πιο δύσκολοι καιροί θα έρθουν στις αρχές του επόμενου έτους. Ε, πρέπει να είμαστε πιο κοντά από ό,τι ποτέ μέχρι τώρα, μέχρι τον Μάη για τις πολιτικές συνοχής. Θα έχουμε εβδομάδα των περιφερειών, αφιέρωση στο, αφιερωθούμε στο μέλλον, αρχές του επόμενου έτους, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα ξεκινήσουμε σε, μέσω μιας διάσκεψης. Πότε στη Σόφια, 9 ε, και 10 Ιανουαρίου, η πρώτη μέρα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, Δευτέρα και Τρίτη, μέρες εργασίας για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο τον Ιανουάριο και θα είμαι εκεί για να προβάλλω τα επιχειρήματα για τη μελλοντική πολιτική συνοχής. Έχουμε 8 και 9 ε, αυτή τη διάσκεψη τον Ιανουάριο. Ελπίζω να είσαστε εκεί, να είναι παρούσα η Επιτροπή σας. Πριν τον Μάιο θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη ορατότητα και εσείς τα κράτη-μέλη σας πρέπει να είσαστε πιο ορατοί να προβάλλετε τις συμμαχίες αυτές της συνοχής, τη συντονίζει η Επιτροπή των Περιφερειών και το Κοινοβούλιο. Τον Μάρτιο γιορτάζουμε 30 χρόνια πολιτικής συνοχής και αυτή τη σημαντική στιγμή μπορούμε να δείξουμε τι έχει επιτευχθεί σε τόσα πολλά κράτη-μέλη στα 30 χρόνια από όταν ετοιμάσαμε αυτό το, το ταμείο που είναι το Ταμείο Αλληλεγγύης Οικονομικής. Διάφορες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κεντρική εκδήλωση είναι 24 Μαρτίου. Σας καλώ όλους να είστε παρόντες. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα που θέσατε μπίπτει στην αρμοδιότητα του κυρίου Ντομπρόφσκης, από ό,τι γνωρίζω, και άλλοι πόροι προέρχονται από τα αποθέματα του Ευρωπαϊκού Υπολογισμού για το ΣΥΕΡΑ. Ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι μια πολύ καλή εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο. Δεν τα ξαναπούμε. Στο Στρασβούργο, έτσι. Για μια ακόμη φορά. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στο Στρασβούργο. Ελπίζω να ολοκληρώσουμε επί του όμνιμπους ε, το, τις εργασίες αποκριστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Ρέτζη. Ελπίζω έτσι να κλείσει καλά το έτος. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Με τα χαρά σας ξαναδούμε. Ολοκληρώνεται το πρώτο τμήμα της συνεδρίασής μας. Θα συνεχίσουμε υπό τη μορφή συντονιστών άνευ διερμηνίας, δυστυχώς λέει ο Πρόεδρος, στα αγγλικά. Εμείς σας ευχόμαστε καλή όρεξη αργότερα.